Guten Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αργήσει η Πρόεδρος και δεν είναι παρόντες οι αντιπρόεδροι, γι' αυτό θα ξεκινήσω εγώ τη συνεδρίαση. Προχωράμε λοιπόν κατευθείαν στην ημερήσια διάταξη. Υποθέτω ότι μπορεί να εγκριθεί ως έχει. Καλώς. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Διερμηνία υπάρχει προς όλες τις γλώσσες εκτός από την Κροατική. Έχουμε επίσης την ανακοίνωση ότι ο κύριος Τιμ Άκερα από το ΕΛΚ έγινε αναπληρωτής ε, στην ε, Επιτροπή μας. Ε, τον καλωσορίζουμε και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μαζί του. Έχουμε επίσης μια ομάδα προσκεκλημένων που θα καταλαβαίνουν πολύ καλά τα γερμανικά μου. Μια ομάδα λοιπόν από εκπροσώπους ε, του, επιμελητηρίου, του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Σαξονίας. Ε, σας καλωσορίζω θερμά στην Επιτροπή μας. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε μια ακρόαση ε, και μία ακόμα ανακοίνωση. 15-18 Μαρτίου η Επιτροπή μας ε, έχει προγραμματίσει αποστολή στην Κοπενχάγη. Κάποια μέλη επισκέφτηκαν την Κοπεχάκη και την πόλη Σλάγκελσε, όπου επικεντρώθηκαν ε, στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. καθώς και με την αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Στα έγγραφά σας θα βρείτε μία σύνοψη αυτής της αποστολής. Φτάνουμε έτσι στο πρώτο θέμα ουσίας της σημερινής συνεδρίασης, που είναι η δημόσια ακρόαση για την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Η ακρόαση αυτή προγραμματίστηκε σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου του 2014. όπου ασχοληθήκαμε με τις πτυχές απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της Ευρω... Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Στόχος είναι η επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής να γίνει μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση. Θέλουμε συμμετοχή των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών. Και γι' αυτό ε, τα συμπεράσματα θα συμπεριληφθούν στην ε, δημόσια διαβούλευση της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Σύντομα θα σας παρουσιάσω τους σημερινούς μας προσκεκλημένους. Στο βαθμό που είναι παρόντες. Αρκετοί από αυτούς επίσης έχουν καθυστερήσει, γι' αυτό αυτό σχεδιάζουμε σήμερα. Ο δόκτωρ Φρανκ Γιούργεν Βάιζε, πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και επικεφαλής της ομοσπονδιακής για την απασχόληση. Δεύτερη προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Φρανσουάζ Ντομποέ. Είναι συντονίστρια της Βέλγικης Υπηρεσίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κυρία Έλεν Νίκρεν προέρχεται από την συνδικαλιστική οργάνωση LO της Σουηδίας και είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής ε, Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ιδιαίτερα για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων. Κατόπιν έχουμε την κυρία Μπάρμπαρα Χέλπερι, αντιπρόεδρο της Κοινωνικής Πλατφόρμας και πρόεδρος της Semester Alliance. Κατόπιν έχουμε τον κύριο Μάουρο Καπέλο, που είναι ελεγκτής της ελεγκτικής αρχής της Υπηρεσίας της Εθνικής Συνοχής της Ιταλίας. Και τέλος έχουμε την κυρία Ντόρτε Άντερσεν, που είναι διευθύντρια ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ε, Ένωση Δανών ε, Εργοδοτών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία και ξεκινάμε την ακρόαση. Ο καθένας έχει 8 λεπτά για να μας παρουσιάσει τους συλλογισμούς του κατόπιν οι συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ε, Δόκτωρα Βάιζα, σας παρακαλώ να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε και εσείς. Εκπροσωπώ τους 28 ε, διοικητές των ε, Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης η πολιτική μας λέει τι πρέπει να γίνει και εμείς είμαστε αρμόδιοι για την αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή. Τρεις λέξεις κλειδιά θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς, μία παρατήρηση όσον αφορά το θεματολόγιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης. Η εργασία, κατά τη γνώμη μας, έχει προτεραιότητα. Καταπολεμούμε έτσι την φτώχεια. Υπάρχουν ε, οι άτυπες μορφές εργασίας, η μερική εργασία για παράδειγμα ή η κακά πληρωμένη εργασία, η οποία όμως παρόλα αυτά είναι προτιμητέα σε σχέση με την ανεργία. Διότι μπορεί να αποτελέσει ε, εισιτήριο για την αγορά εργασίας η εργασία δεν είναι ένα συγκεκριμένο όγκο ο οποίο μοιράζεται. Όσο περισσότεροι δουλεύουν, τόσο περισσότερε θέσει απασχόληση δημιουργούνται. Και γι' αυτό βλέπουμε σε κάποιε χώρε συνεχή αύξηση τη απασχόληση. Και τέλο, όσον αφορά την πολιτική απασχόληση, μα φαίνεται όλο και πιο σημαντικό όχι μόνο να καταπολεμήσουμε την ανεργία, αλλά να υπάρχουν και μέτρα πρόληψης ε, κατά της ανεργίας, για παράδειγμα η καλή συνεργασία με το εκπαιδευτικό σύστημα. Χρειαζόμαστε επαγγελματοποίηση των υπηρεσιών αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει νόημα να επενδύουμε σε κακές δομές. Υπάρχει μία υπόθεση όσον αφορά τα χαμηλά πρότυπα. Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός ήδη στο σχολείο, η διαφάνεια όσον αφορά τις θέσεις εργασίας απέναντι στους ετούντες, στρατηγικές επιγραμμικές, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι άνθρωποι αλλά και η προσωπική παροχή συμβουλών είναι σημαντικά. Θέλουμε λοιπόν ένα ενεργό πρόγραμμα απασχόλησης, περιφερειακό, ώστε να λαμβάνει διαφορετική μορφή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας και πιστεύουμε ότι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα πρέπει να κατέχουν ηγετική θέση στο θέμα αυτό. Επίσης, απαιτείται συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με όλους τους εταίρους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση κλπ. Τρίτον, πιστεύουμε ότι η Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 αποτελεί κατάλληλο μέσο για να υπάρχει συνεχής βελτίωση. Είναι αλήθεια ότι οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί δεν έχουν επιτευχθεί. Είναι όμως λάθος να πιστεύει κανείς ότι όλοι οι στόχοι που διατυπώνονται στην αρχή του έτους θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί στο τέλος του έτους. Η διατύπωση των στόχων ε, έχει να κάνει με το τι απομένει να γίνει, τι δεν έχει να γίνει, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Και η εγγύηση για την νεολαία αποτελεί καλό παράδειγμα των στοιχείων που συγκρίνουμε μεταξύ των 28 κρατών μελών. Τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, τι μάθαμε από όλα αυτά. Και υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις. οι υπηρεσίες απασχόλησης δημοσίου δικαίου εργάζονται σύμφωνα με τον όρο, με την έννοια του bench learning. Δηλαδή έχουμε δείκτες, συγκρίνουμε τα ευρήματα μεταξύ τους, δημοσιεύουμε τα καλά παραδείγματα και έτσι πετυχαίνουμε να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Τα κακά παραδείγματα τα κρατάμε για τον εαυτό μας, για να μην κατηγορούμε κανέναν. Και στόχος είναι καθένα από τα 28 κράτη-μέλη να βελτιώνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην Γερμανία από το 2005 10 χρόνια χρειάστηκαν ώστε από μια όχι πολύ καλή θέση όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, καταφέραμε να κατέχουμε πολύ καλύτερη θέση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μας φαίνεται ότι αυτό είναι καλό στοιχείο και ε, γι' αυτό θέλουμε να σας εθαρρύνουμε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Βάισε. Η κυρία Ντεμποέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω σε 8 λεπτά να σας πω την ουσία αυτών που πρέπει να πω. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η δημόσια υπηρεσία από το Πέλιο δεν είναι γνωστή. Εμείς πρέπει να αποτιμήσουμε την ε, αποδοτικότητα του ε, πρωτογενούς δικαίου για την αντιμετώπιση της ε, φτώχειας. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρωτογενές ε, δίκαιο το οποίο να μπορεί να αντισταθεί στη φτώχεια. Μιλάμε για τον τομέα της υγείας, μιλάμε για το προσδόκιμο ζωής, για μειονεκτούσες καταστάσεις και ξέρουμε ότι η χαρακτηριστική ασθένεια της φτώχειας ε, είναι ακριβώς ε, η μειωμένη αντίσταση στις ασθένειες. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, να ορίσουμε ένα πλαίσιο αποτίμησης για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που ζουν σε κατάσταση φτώχειας. Θα σας εξηγήσω τη θέση μου τη θέση μας και θα σας πω τι είδαμε στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Μετά θα μιλήσω για τα αποτελέσματα και για το μέλλον. τα ενδυνάμει ενδιαφέροντά μας σχετίζονται με μια εγκάρσια προσέγγιση γιατί υπάρχει ε, το θέμα της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πραγματικότητας. Η οικονομική ανάπτυξη κάθε αυτή δεν μειώνει αυτόματα τη φτώχεια και τις ανισότητες. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε αυτά τα δύο στοιχεία για να φτάσουμε στη σύγκληση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου για όλους. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι θετικό στην Στρατηγική Ευρώπη 2020, σχετίζεται με την καταπολέμηση της φτώχειας κάθε αυτή. Θα επανέλθω σε αυτό για να δούμε ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί. Θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Τέλος, το τρίτο θετικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει σωρία δικτών που χρησιμοποιούνται για να δούμε την πρόοδο ή τις παλινοδίες στον τομέα της φτώχειας και βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί δείκτες που χρησιμοποιούμε και βλέπουμε πολλές ομάδες φτώχειας. Δηλαδή, με τρεις δείκτες ορίζουμε όλες τις ομάδες φτώχειας και βλέπουμε ότι υπάρχουν και κοινοί τόποι. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, ξέρετε ότι έχουμε πολύ λίγα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, γιατί όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η ίδια η Επιτροπή λέει ότι δεν θα μπορέσει σύντομα η Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, τα αριθμητικά στοιχεία υποτιμούν τον αριθμό των φτωχών. Αυτό το βλέπουμε και στο Βέλγιο, γιατί οι δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη τις κατηγορίες που βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση όπως τους άστεγους, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στα δείγματα της έρευνας. Προωθήσαμε λοιπόν ένα ε, πλαίσιο έρευνας έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και τους αστέγους στη, στο δείγμα, στα δείγματα που χρησιμοποιούμε για να προσπαθήσουμε ώστε η έρευνα να λάβει υπόψη όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρξουν αποδοτικά συστήματα προστασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Βλέπουμε ότι η οικονομική πτυχή αναπτύχθηκε κατά ε, της πτυχής του κοινωνικού αποκλεισμού. Λάβαμε υπόψη στους μισθούς και στα διάφορα ευεργετήματα χωρίς να λάβουμε υπόψη την κοινωνική προστασία γενικότερα. Ε, δηλαδή αυξάνονται η, αυξάνεται η εργασία αλλά δεν σημαίνει ότι και η ποιότητα ε, ζωής και διαβίωσης των φτωχών ε, βελτιώνεται γιατί υπάρχουν ευάλωτες κατηγορίες και σίγουρα όταν έχουμε να κάνουμε με μία ε, εργασία με σύμβαση, στη συνέχεια μπορεί κανείς να έχει σύμβαση αορίστου χρόνου, αν έχει αρκετά προσόντα. Ενώ αν δεν έχει πολλές δεξιότητες, όχι. Στο μέλλον θέλουμε να φτάσουμε στην πρώτη ε, φιλοδοξία, δηλαδή στην ε, εγκάρσια προσέγγιση και στην οριζόντια κοινωνική ρήτρα. Υπάρχουν μέσα, όπως για παράδειγμα, το, η, η η οριζόντια κοινωνική ρήτρα που προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο μέσο είναι να έχουμε αριθμητικά στοιχεία της στρατηγικής 2020 μέσα στα πλαίσια μιας εγκάρσιας προσέγγισης. Είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε σε στοιχεία για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλείσμου. Όταν ε, ληφθούν μέτρα, ίσως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα μέσα στα πλαίσια ε, μιας εγκάρσιας προσέγγισης και συνοδευτικής. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα ετήσια σχέδια μεταρρύθμισης που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη στις ευρωπαϊκές αρχές και την ε, έκθεση για την ε, κοινωνική αντιμετώπιση του ζητήματος που έχει μεγάλη σημασία τουλάχιστον στη χώρα μου. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η εργασία, η θέση εργασίας, αλλά Ποιοτικέ θέσει εργασία που να σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, γιατί ξέρουμε ότι όσοι, όσοι έχουν λιγότερα προσόντα απομακρύνονται από την αγορά εργασία για μακρύ χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να υπάρχει μία κοινωνική προστασία υπέρ των πλέον αδυνάμων και αυτό αφορά ε, και μία αρχή αιρεσιμότητας ως προς τα δικαιώματα θα πρέπει να υπάρχει μία δραστηριοποίηση με τα τρία στοιχεία, ε, αξιοπρεπής μισθός, αγορά εργασίας και ανοιχτή ε, αγορά και αντιμετώπιση. Σε καιρούς κρίσης ε, η κοινωνική προστασία πληρώνει τα σπασμένα, όμως πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα και μία επένδυση για το μέλλον. Και η τέταρτη προτεραιότητα είναι η συμμετοχή καθεαυτή, διότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να σχετίζονται με συγκεκριμένα ε, επαγγέλματα και υπηρεσίες, μία επανεπεξεργασία δηλαδή, η οποία θα γίνεται από τη βάση και δεν θα επιβάλλεται εκ των άνω. ένα δεύτερο στοιχείο και είναι και το τελευταίο, να συμπληρώσουμε τα αριθμητικά στοιχεία με ποιοτικούς ε, προσδιορισμούς. Τα αριθμητικά στοιχεία θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι αναγκαία, αλλά πέρα από τον προσήκοντα χαρακτήρα τους, ε, θεωρούμε ότι τα αριθμητικά στοιχεία για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, μπορούν να εμπεριέχουν κινδύνους, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη τους πιο φτωχούς, όπου θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη φτώχεια. Ίσως φτάνουμε στο στόχο, αλλά υπάρχει μεγάλη ανισότητα, ενώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνική συνοχή. Αριθμητικά στοιχεία και στοχοθέτηση. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί θέλουμε ένα μέρος, ένα κοινωνικό στρώμα να βγει από την φτώχεια και αυτό ακριβώς σας εξήγησα όταν σας μίλησα για το στόχο της μείωσης ε, της φτώχειας. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση του 2020, αν έχουμε πέντε ανέργους, αν είχαμε πέντε ανέργους γύρω από ένα τραπέζι, ο ένας πια δεν θα είναι φτωχός και άνεργος μετά από πέντε χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο ποιοτική προσέγγιση, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε πώς και με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να βγει από τη φτώχεια ε, πραγματικά και όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της ε, στοχοθέτησης και μετά να, ξαναβρεθεί, να ξαναβρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στη φτώχεια. Ευχαριστούμε. Κυρία Ντεμπόε, είσαστε συντονίστρια της Βελγικής Υπηρεσίας της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο επόμενος, η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Νίγκρεν, που εκπροσωπεί την ε, LO, την, ε, τα σουηδικά συνδικάτα και ασχολείται με θέματα κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα ως προς τα εργασιακά σχήματα. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σουηδικά, εφόσον έχω τη δυνατότητα. Εκπροσωπώ τη συνδικαλιστική οργάνωση LO, μία από τις τρεις κεντρικές νομοσπονδίες στη Σουηδία. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε λοιπόν τρεις κεντρικές συνομοσπονδίες. Στην LO έχουμε τους εργαζομένους, η ε, TCO και η ΣΑΚΟ εκπροσωπούν ε, τους πανεπιστημιακούς συνεργαζόμαστε όμως ε, πολύ συχνά και ειδικά για ευρωπαϊκά θέματα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι στην Σουηδία οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με τους ε, κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της στρατηγικής ε, Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 λειτουργεί πολύ καλά. Φυσικά μπορεί να βελτιωθεί. Ε, αλλά βλέπουμε ότι ακούγονται οι απόψεις με σεβασμό. Οι τρεις αυτές συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουμε στη Σουηδία η ΕΛΟ, και η ΣΑΚΟ. Ε, ανήκουν και οι τρεις στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ε, στην ΕΛΟ συμμετέχουν 14 ε, οργανώσεις, ενώ οι άλλες εκπροσωπούν δημοσίους, υψηλούς δημοσίους αξιωματούχους και πανεπιστημιακούς. Κατά καιρού έχουμε διαφορετικέ προτεραιότητε. παρόλα αυτά, όσον αφορά τα θέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Οι εργοδότε εκπροσωπούνται στην Σουηδία μέσω ε, μεγάλων οργανώσεων που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Έχει ξεκινήσει διαβούλευση σε τακτική βάση με τους κοινωνικούς εταίρους στη Σουηδία. Μία φορά το χρόνο ε, προσκαλούνται ε, οι εταίροι ε, σε υψηλό επίπεδο και κατά καιρού προσκαλούνται και οι ειδικοί για διαβουλεύσεις. δημόσιοι υπάλληλοι από διάφορα υπουργεία, συνήθως είναι παρόντα στις διαβουλεύσεις, ακούνε τις απόψεις μας και απαντούν σε ερωτήσεις. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών κάθε χρόνο υποβάλλουν γραπτή συνεισφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Επίσης ε, συμβάλλουν και εθελοντικές οργανώσεις. Να προχωρήσουμε τώρα όμως στην αξιολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ε, αν επικεντρωθούμε στους στόχους για την απασχόληση και την καταπολέμηση της στόχιας, είναι θετικό ότι υπάρχουν ως βασικές αρχές στην ευρωπαϊκή και την ε, εθνική πολιτική. Εφόσον όμως απέχουμε πολύ από την επίτευξη των στόχων, είναι σαφές ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η στρατηγική θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τι μπορεί να βελτιωθεί. Η κοινωνική στόχοι στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι καλή και σημαντική. Διαπιστώνουμε όμως ότι ο, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και οι μη δεσμευτικοί δείκτες δεν αρκούν ώστε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση λείπει μία σαφής κοινωνική ατζέντα, ένα κοινωνικό θεματολόγιο. Οι 26 εκατομμύρια ε, ανέργους έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 20 εκατομμύρια ε, που ζουν κάτω από το ε, όριο της φτώχειας. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων έχει διατυπώσει 10 βασικούς στόχους για αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Να επιτευχθούν οι ε, προσδοκίες, να εκπληρωθούν οι προσδοκίες ε, με αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Επενδύσεις ε, στην ΕΦΗ e e και βιώσιμη ανάπτυξη. Να κάνουμε τώρα βήματα αποφασιστικά. Να δώσουμε τέλος στην λιτότητα, να συμμετέχουν οι ε, ε, εταίροι σε μεγαλύτερο βαθμό στην ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει να έχουμε προληπτικά και διορθωτικά μέτρα. Η στρατηγική θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες πολιτικές προκλήσεις, ιδιαίτερα ένα κοινωνικό θεματολόγιο. Να μην επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να κατακαιρματίζουν τους ε, φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους σε λιγότερο φιλόδοξους εθνικούς στόχους και να έχουμε μια πλουραλιστική κοινωνική συζήτηση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία ε, Χέλφρις, αντιπρόεδρο της Κοινωνικής Πλατφόρμας. Παρακαλώ. Yes, thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πλατφόρμας και της Ένωσης για την αηφόρο προστασία των εργαζομένων και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σε αυτήν εδώ τη συνάντηση την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Η αναθεώρηση αυτής της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και είναι πολύ θετικό για μας που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προσεκάλεσε και μη κυβερνητικέ οργανώσεις για αυτό το στόχο. Η κοινωνία των πολιτών περίμενε ε, με αγωνία και ενδιαφέρον θα έλεγα την ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση και η καθυστέρηση μέχρι το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του 16 είναι κάτι το οποίο μας απαγοήτευσε και είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέπειες και για την ίδια την αξιολόγηση. Τώρα λίγα λόγια για την κοινωνική πλατφόρμα. Αποτελείται από 46 ε, μίζονες μικιό που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα σε επίπεδο κρατών μελών. η Ένωση για ένα σοσιαλδημοκρατικό και αηφόρο εξάμεινο. Συνεργάζονται έτσι ώστε όλες οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα από το 2011 να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πρόοδο γύρω από το εξάμεινο αυτό σε σχέση με τους λεγόμενους κοινωνικούς στόχους. Θα μπορούσα να πω περισσότερα. Η πλατφόρμα είναι λίγο ευρύτερη σε σχέση με τα μέλη της και θα έχω πάρει το λόγο σαν αντιπρόεδρος ακριβώς της social platform, της κοινωνικής πλατφόρμας. Εμείς παρακολουθούμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ασκήσαμε κριτική ε, στις υποσχέσεις που είχαν δοθεί και στις ε, εφαρμοσμένες πολιτικές. Βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε 5 εκατομμύρια περισσότερους πτωχούς από ότι το 2010 έχουν μειωθεί τα επίπεδα απασχόλησης, δεν ξεπερνούν το 68% και είναι ακόμα χαμηλότερα για τις γυναίκες και για συγκεκριμένους κοινωνικούς, κοινωνικές κατηγορίες. Υπάρχει επίσης πάντα μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις αμοιβέ ανδρών γυναικών 39% ε, διαφορά στις συντάξεις και στο Λουξεμβούργο 47% και την Γερμανία 44%. Τρομακτικές διαφορές δηλαδή, οι οποίες αποδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα ε, και την αστοχία γενικά της προσπάθειας γύρω από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Συνεπώς η αναθεώρηση είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Εμείς προσπαθούμε να εξετάσουμε τους στόχους που είχαν τεθεί από το 11. Είδαμε ότι δίδεται πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις οικονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές κυρίως. Αυτό σημαίνει ότι οι συστάσεις χώρα έχουν σαν στόχο τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη μείωση γενικότερα των δημοσίων δαπανών. Συνεπώς δεν υπάρχει συνεκτικότητα ανάμεσα στους στόχους και, την και τα μέτρα επιδίωξης των στόχων αυτών. Και αυτό γεννά όλο και περισσότερη φτώχεια. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πλατφόρμα έχει τρεις μείζονες συστάσεις εδώ. Η πρώτη είναι η διασφάλιση της συνεκτικότητας των πολιτικών και της διαφάνειας των διαδικασιών. Απαιτείται η αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής Ευρώπη 2020 και της διαδικασίας του εξαμήνου, έτσι ώστε τα μέσα και οι πολιτικές να ανήκουν σε μια ενιαία στρατηγική και να λειτουργούν περισσότερο διαφανώς ε, μέσω των διαδικασιών που συνοδεύουν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η δεύτερη σύσταση είναι η διασφάλιση προόδου στον τομέα των κοινωνικών στόχων. Αυτά τα είπε και ο προλαλής σας. στόχος είναι η μείωση της ένδυας, του κοινωνικού αποκλεισμού, να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα ανισότητας και στον τομέα της ανεργίας και όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης και όλα αυτά στα πλαίσια των στόχων της Ευρώπης 2020 και η τρίτη σύσταση έχει σχέση με τους εμπλεκομένους και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και σε εθνικό επίπεδο και εν μέρη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κοινωνία των πολιτών δεν εμπλέκεται με τον κατάλληλο τρόπο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών του εξαμήνου. Και τα εθνικά προγράμματα και τα κοινωνικά προγράμματα δεν αξιολογούνται σωστά και η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών είναι ανεπαρκής και πολλές φορές δεν χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα, υπάρχει μια πρώτη συνάντηση και πέραν τούτου ουδέν και καμία μορφή συντονισμού της κοινωνίας των πολιτών με τις εθνικές αρχές. Τώρα σε σχέση με τη διαφάνεια των πολιτικών είπαμε ότι ο κοινωνικός παράγων έχει χάσει σε σχέση με τον οικονομικό παράγοντα και σε επίπεδο εξαμήνου απαιτείται μία επανεξισορρόπηση. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν στα πλαίσια της αναθεώρησης της Ευρώπης 2020. Απαιτείται να υπάρξει επίσης και μία μορφή εκ των υστέρων των οικονομικών, κοινωνικών και φορολογικών πολιτικών, αλλά και εκ των προτέρων μία αξιολόγηση σε επίπεδο διαφοράς φύλων και κυρίως στον τομέα της διαφοράς των αμοιβών. Απαιτούνται επίσης συγκεκριμένες δράσεις σε όλους τους στόχους τους κοινωνικούς στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης και ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη περισσότερα στοιχεία για την καταγραφή της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι εξαιρούνται οι χώρες κάτω από τρόικα από την εφαρμογή των CSR, των CSR όπως οι υπόλοιπες χώρες. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και για την, το mainstreaming της ισότητας των φύλων και για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε να υπάρχει μια ετήσια έκθεση, τακτική έκθεση στα πλαίσια ακριβώς της αξιολόγησης και παρακολούθησης των εξελίξεων. Ο Πίνακα στόχων, το scoreboard, έχει ακολουθηθεί και παρακολουθηθεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς θα θέλαμε να συμπληρωθεί και από περαιτέρω δράσεις διορθωτικές όταν βλέπουμε ότι ορισμένοι τομείς διαφεύγουν ελέγχου και δεν επιτυγχάνουμε τους κοινωνικούς στόχους. Ο πίνακας αυτών στόχων, το στοχολόγιο αν θέλετε, έχει να κερδίσει από μια πιο αναλυτική ανάλυση και των ακραίων μορφών ένδυας. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους δείκτες που χρησιμοποιούμε και να τους καταστήσουμε πιο αποκαλυπτικούς για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ζητάμε λοιπόν για ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Θέλουμε οι στόχοι να κατανεμηθούν ανά ομάδα, ανά θεματολογία, ανά φύλλο. Όταν λέω θεματολογία εννοώ τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση. Θέλουμε επίσης μια σωστή εφαρμογή του κοινωνικού πακέτου στον τομέα της καταπολέμησης του φαινομένου των αστέγων ε, όπως επίσης και την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Για το τρίτο θέμα τώρα, τον, την εμπλοκή ε, των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων, εμείς σαν κοινωνία των πολιτών παρακολουθούμε από κοντά τις διαδικασίες, μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε πετύχει τον λεγόμενο διαρθρωτικό διάλογο με τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές πάνω στις παρατηρήσεις μας. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, εκεί έχουν βελτιωθεί οι επαφές ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τα κοινωνικά και οικονομικά υπουργεία. Σε άλλες χώρες κάτι τέτοιο όμως δεν λειτουργεί και ο διάλογος είναι μόνο κατόνομα πραγματικός. Απαιτείται λοιπόν κατευθύνση σωστή έτσι ώστε να διαρθρωθεί ο συγκεκριμένος διάλογος και να εφαρμοστεί και η αρχή της εταιρικότητας στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου. Μια τελική παρατήρηση τώρα οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα μέλη της κοινωνικής πλατφόρμας διαπιστώνοντας τις αλλαγές στις συστάσεις αναχώρα τον τελευταίο καιρό και τις παρατηρήσεις ε, που γίνονται γύρω από τη συνέχιση ε, της ε, λιτότητας υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις ειδικέ γι' αυτό που έχουν μειωθεί από 12 σε 6 και βλέπουμε ότι στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα και όχι η αναζήτηση δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Και μία ακόμα τελευταία τρίτη φορά λέξη, ε, οι συστάσεις αναχώρα μέχρι τώρα δεν δείχνουν μια ενιαία στρατηγική. Διαρωτώμεθα λοιπόν γιατί η μεθοδολογία ακριβώς αυτής της διατύπωσης αυτών των εκθέσεων τι νόημα έχει εάν δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να τη συνδυάσουμε. Thank Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάουρο Καπέλο, δημοσιονομικός ελεγκτής από την Υπηρεσία Εθνικής Συνοχής της Ιταλικής Δημοκρατίας. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Κύριοι βουλευτές, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Θα μιλήσω για την αναθεώρηση της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θα ασχοληθώ με την κατάρτιση και την εκπαίδευση και τις συγκεκριμένες πολιτικές για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σχετίζονται με τη δυνατότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες να αρχίσουν να σκέφτονται κατά καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να ασχοληθούμε με την, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον άνθρωπο με την απόφαση 1350 του 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι το 2009 είναι έτος καινοτομίας και δημιουργικότητας και υπήρχαν και κατευθυντήριες γραμμές μέσα σε αυτή την απόφαση στην ε, σύσταση 962 του 2009 μιλήσαμε ακριβώς για διαβίου μάθηση. Ε, μιλούσαμε για ένα πρόγραμμα ε, «Μαθαίνω να εκπαιδεύομαι». Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιες είναι οι τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2014 ήταν έτος που αφιερώθηκε στον εγκέφαλο, στις εγκεφαλικές διεργασίες και ασχοληθήκαμε φυσικά και με θέματα νευρολογικών και ψυχολογικών ασθενειών, καθώς και με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Η πρότασή μου, πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 να μιλήσουμε για μια πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο «Ανακαλύπτοντας τη σκέψη», «Ανακαλύπτοντας τον εγκέφαλο», που σχετίζεται με τους νέους Ευρωπαίους που ασχολούνται με θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Να τους δείξουμε πώς ε, λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, όπως ε, μάθαμε από την επιστήμη και ποιες είναι οι τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκμάθησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δυνατότητα συσχετισμού που είναι η βάση της ε, γνωσιακής διεργασίας. Κύριοι βουλευτές, σας προτείνω να δούμε πώς μπορούμε να επαυξήσουμε αυτές τις γνώσεις ως προς τις ε, διανοητικές διεργασίες. Θα προωθηθούν συγκεκριμένα σεμινάρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την επαγγελματική κατάρτιση μεταξύ άλλων και να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι τεχνικές ε, της γνωσιακής διεργασίας μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας διαχείρισης. Μιλώ για το mind mapping και για το brainstorming θα είχε μεγάλη σημασία στα πλαίσια αυτά να προωθήσουμε εκστρατείες με συγκεκριμένα ε, μηνύματα, στοχοθετημένα και να προτείνουμε και μελέτες σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών, αλλά και ευρωπαϊκών. Σας προτείνω να προωθήσουμε στα πλαίσια των ε, διαχειριστικών προγραμμάτων και των λειτουργικών προγραμμάτων να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, τεχνικές απομνημόνευσης και πώς μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό το, το γνωσιακό πλαίσιο στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη λογοτεχνία ακόμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε την χαρτογράφηση του εγκεφάλου και του νου για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, απόφαση που έχουμε και τις ε, συστάσεις που ακολουθούν. Τέλος, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο ε, είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της γνώσης που να απευθύνεται σε όλους τους νέους, τους νέους Ευρωπαίους, ακολουθώντας ε, αυτό το, αυτή τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου μυαλού. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο αυτές οι τεχνικές μας έχουν βοηθήσει για την καλύτερη προώθηση των γνώσεων αλλά και την ποιότητα εκμάθησης. Προτείνω αυτές τις δραστηριότητες γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία σωστή διεργασία εκμάθησης και αλφαβητισμού μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Κάποιος είπε ότι το μυαλό ε, είναι σαν ένα αλεξίπτωτο, λειτουργεί καλά μόνο όταν ανοίξει. Για να ανοίξει λοιπόν ένα αλεξίπτωτο θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να έχει το θάρρος να το ανοίξει. Γι' αυτό εσείς που είσαστε η κινητήριος δύναμη της Ευρώπης θα ήθελα να ε, προωθήσετε αυτό το άνοιγμα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε λέτε να είμαστε παράτολμοι με άλλα λόγια. Η κυρία Ντόρτε Άντερσον έχει τώρα το λόγο. Ποιος είδαμε. Και είναι υπεύθυνη ε, από πλευράς ε, των εργοδοτών δηλαδή, στα πλαίσια της ε, ε Συνομοσπονδίας Εργοδοτών. Έχετε το λόγο. Μεγαλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Εκπροσωπώ την Ένωση Εργοδοτών της Δανίας. Εκπροσωπούμε περίπου 24.000 δανέζικες εταιρείες. Κάτι που αντιπροσωπεύει περίπου το μισό των δανών απασχολούμενων. θα προσπαθήσω να σας δώσω τρεις βασικές προτάσεις ε, σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είναι λίγο δύσκολο να είναι κανείς ο τελευταίος ομιλητής ε, μετά από πέντε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ. Οι τρεις προτάσεις μας είναι λοιπόν. Πρώτον, διατηρήστε τον στόχο της απασχόλησης. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εξετάζεται σε πιο ευρύ χρονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να, δηλαδή να έχουμε κατά νου και τι μορφή θα έχει ο κόσμος μετά το 2020. Η άλλη πρόταση αναφέρθηκε ήδη, έχει να κάνει με το benchmarking. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ καλύτεροι σε αυτό που κάποιοι αποκαλούν bench learning, δηλαδή υψηλότερη ποιότητα στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση καθώς ε, και στις ε, ανταλλαγές όσον αφορά την εκπαίδευση. Τέλος, μία έκκληση μάλλον περισσότερο προς τα κράτη-μέλη. Να συμμετέχουν στις εργασίες αυτές πολύ περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι. Πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν σήμερα στην Ευρώπη και στο εγγύς μέλλον. Κάποιοι θα πούν ότι φαίνονται κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εγώ όμως ε, θεωρώ ότι ε, η ανάπτυξη πραγματοποιείται αλλού εκτός Ευρώπης και ότι η Ευρώπη γυράσκει. Μία μικρή χώρα όπως είναι η Δανία εξαρτάται απολύτως από την ανάπτυξη της Δανίας. Μεγάλα μέρη των εξαγωγών μας ε, έχουν προορισμό την Ευρώπη. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι τα πράγματα πάνε καλά στη Δανία. Έχουμε απασχόληση ποσοστό απασχόλησης 80%, αλλά εξαρτώμεθα από το πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή δεν πάνε πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε τον στόχο της ε, απασχόλησης, θα πρέπει όμως να έχουμε και έναν στόχο ανάπτυξης. Και θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα σε 5, 10, 20 χρόνια ε, για να λάβουμε υπόψη μας τις δημογραφικές εξελίξεις θα πρέπει να εξετάσουμε και την προσφορά εργατικού δυναμικού στο μέλλον. Θα πρέπει περισσότεροι να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, να ξεφύγουν ε, από ε, τα κοινωνικά επιδόματα αρκετές επιχειρήσεις ψάχνουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουν, ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετοί άνεργοι. Σε άλλα μέρη της Ευρώπης θα πρέπει να ενταχθούν περισσότερο οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε και με αυτό. Σημαντικός τομέας λοιπόν είναι οι νέοι και η εκπαίδευση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται πολύ η επαγγελματική κατάρτιση όπως και το work-based learning, η πρακτική άσκηση. Στον ιδιωτικό τομέα το εργατικό δυναμικό αυτό είναι ο πυρήνας για πολλές επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και πιστεύω ότι αυτό ισχύει και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ε, για να το πω κάπως ε, σκληρά, εκπαιδεύουμε τους νέους να είναι άνεργοι. Κάτι που έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση, στην νέα αναθεωρημένη στρατηγική Ευρώπη 2020. Το άλλο μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω έχει να κάνει με το bench learning. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό πολύ περισσότερο για να πετύχουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να έχουμε αγορές εργασίας που να λειτουργούν σωστά, ώστε να έχουμε και ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης και υψηλότερης ποιότητας θέσεις απασχόλησης, ώστε οι επιχειρήσεις να ξαναρχίσουν να επενδύουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μέσα ώστε στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη να έχουμε υψηλότερη ποιότητα. Και μία ακόμα πρόταση. Να έχουμε ένα benchmark όσον αφορά τις ανταλλαγές ε, στο... Ε, στις ανταλλαγές ε, στο σύστημα εκπαίδευσης. Το τελευταίο μου μήνυμα έχει να κάνει περισσότερο με τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Εμείς είμαστε οργάνωση εργοδοτών. Μαζί με άλλες 30 οργανώσεις, ε, κοινωνικούς εταίρους ε, και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, συμμετέχουμε σε ένα φόρουμ πολλαπλών ενδιαφερομένων. Αυτό δεν δημιουργεί αίσθημα οικειοποίησης της στρατηγικής 2020. Ακόμα λοιπόν και αν έχουμε εξελίξεις με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την και το σχέδιο Juncker θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε αίσθημα οικειοποίησης και σε εθνικό επίπεδο επίσης. Οι κοινωνικοί εταίροι στη Δανία ζήτησαν από την κυβέρνηση να υπάρχει πιο στενή συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, διότι εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Ίσως λοιπόν μερικές φορές να μπορούμε να καταλήξουμε και σε κοινέ λύσεις. Η τελευταία μου πρόταση είναι κάτι που ίσως να έχει ξεχαστεί κάπως. Που θα είναι χρήσιμο ώστε οι στόχοι και οι εργασίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωση 2020 να γίνει πιο αποτελεσματική. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε δεσμευτικούς στόχους, να έχουμε εθνικά, εθνικές συμβάσεις μεταρρύθμισης. Αυτό συζητήθηκε πριν κάνα δύο χρόνια, ξεχάστηκε όμως μετά, απορρίφθηκε τότε. Ίσως όμως θα πρέπει να το ξαναεξετάσουμε, δηλαδή πώς μπορούν οι εργασίες να γίνουν πιο δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη. Θα κλείσω εδώ. Ε, και προσβλέπω στην καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις έξι ενδιαφέρουσες αυτές παρεμβάσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές και τους εκπροσώπους, αναπληρωτές τους. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Σούλτσε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Από πλευράς του ΕΛΚ σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι αυτά που μας παρουσιάσατε ήταν όχι μόνο πολύ ενδιαφέροντα, αλλά αξίζει τον κόπο να τα σκεφτούμε και στη συνέχεια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί τη βασικότερη προτεραιότητά μας. Υπάρχουν διάφορες μορφές απασχόλησης, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς δουλειά. Ακόμα και αν η θέση απασχόλησης ε, δεν ανταποκρίνεται στις δεξιότητες ή δεν είναι πολύ καλοπληρωμένη, είναι πολύ σημαντική ως σημείο εκκίνησης. Και σημαντικό είναι αυτό που ακούσαμε ότι η εργασία δημιουργεί εργασία. Δηλαδή ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης ε, δεν είναι συγκεκριμένος. Επίσης ε, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε την καινοτομία σημαντικό για μας είναι το θέμα της δημογραφικής εξέλιξης. όχι μόνο για μένα που είμαι Γερμανός είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα της απασχόλησης ηλικιωμένων, της απασχόλησης γυναικών, της βελτίωσης της διαβίου εκμάθησης και της διασυνοριακής απασχόλησης. Πολύ σημαντικό θεωρώ επίσης ότι είναι το θέμα των συστάσεων αναχώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει τα εθνικά σχέδια μεταρρύθμισης επίσης ε, να έχουν κεντρικό ρόλο. Δεν έχω πολύ χρόνο, θα είχα κατά τα άλλα πολλά να πω. Να αφήσω το λόγο λοιπόν στους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Στάινροκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι μας παρουσίασαν σημαντικούς ε, συλλογισμούς και θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Μπορεί να μην έχω πιστεί απόλυτα για όλα όσα είπατε, αλλά όπως είπε ο συνάδελφος, θα πρέπει να έχει προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σημαντικό όμως για μας είναι να μην είναι οποιασδήποτε θέση απασχόλησης, θα πρέπει να είναι καλής ποιότητος. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω την πρώτη μου ερώτηση προς τον δόκτορα Βάιζε. Στο Χάφεν είχαμε μία έρευνα σχετικά με τις διάφορες μορφές απασχόλησης και διαπιστώσαμε ότι πολύ λίγοι καταλήγουν σε θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας από τις πιο επισφαλείς μορφές. Στα πολλά χρόνια από τότε, που έχουν περάσει από τότε μου φαίνεται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κιόλα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο δεσμευτική θα πρέπει να είναι η στόχη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θέλαμε 20 εκατομμύρια λιγότερους στοχούς. Βλέπουμε όμως ότι έκτοτε έχουμε 7 εκατομμύρια περισσότερους. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μάθει μέχρι τώρα ότι χρειαζόμαστε ε, δεσμευτικούς στόχους. Κυρία Ντεμποέ, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε στον διάλογο τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, διότι είπατε ότι ο διάλογος είναι πολύ σημαντικό μέσο. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επίσης, προς όλους τους ομιλητές μας θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση. Συζητάμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά πέρα από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν να σκεφτούν τι άλλο να κάνουν. Έχετε προτάσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την Ευρώπη να πετύχει τους στόχους της. Θα ενδιέφερε να ακούσω και τις διάφορες απόψεις που υπάρχουν. Ε, ξεπέρασα και εγώ το μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκινγκ από την ομάδα ALDE. Έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Έφτασα κάπως αργά, αλλά άκουσα τις περισσότερες. Ακούγοντας αυτά που είπατε σήμερα, φαίνεται ότι υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Υπάρχει έλλειψη ε, συνοχής και αυτό που κάνουμε είναι ε, να μην συνδέουμε τα πράγματα μεταξύ τους. Κάτι άλλο που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αποτιμήσουμε τη συνολική προοπτική και όχι να έχουμε μια κερμα... κατακαιρματισμένη ε, προοπτική. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση για να μπορέσουμε να εργαζόμαστε αποδοτικά όταν μιλάμε για τη στρατηγική 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ε, μία συνολική αποτίμηση. Άκουσα από συναδέλφους ότι υπάρχει καθυστέρηση και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιες είναι οι, εθνικές ε, αποτιμήσεις και μεταρρυθμίσεις. Έχουμε ένα βαθμολόγιο των ε, κοινωνικών δικτών αλλά δεν υπάρχει σωστή διορθωτική δράση που χρησιμοποιούμε όταν οι δείκτες αυτοί χτυπήσουν κόκκινο. Θα ήθελα την άποψή σας γιατί οι δείκτες υπάρχουν πολύ συχνά δεν είμαστε σίγουροι για το κατά πόσο ανταποκρίνονται τα κράτη-μέλη, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν υπάρχει κάτι που τους ε, υποκινεί για να φτάσουν σε αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός κίνησης ή όθησης έτσι ώστε να προωθηθεί διορθωτική δράση. Επίσης δεν υπάρχει μία συνδεσιμότητα. Αν δείτε τα διάφορα προγράμματα, το Easy Program, το ε, κοινωνικό σύστημα συντονισμού, η διαδικασία εξαμήνου, το επενδυτικό πρόγραμμα εξαμήνου, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ τους. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Και έχω κι άλλες ε, τρεις ε, παρατηρήσεις. Ακούσαμε για την εργασία και την αξιοπρεπή εργασία. Αυτός ο όρος μου αρέσει διότι τον έχει προσδιορίσει τον όρο αυτό και ο ΔΟΕ. Μία εργασία είναι εργασία, είναι το πρώτο κλιμάκιο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη ακόμα εργασία. Α, έχω υπερβεί το χρόνο. Α, έξι. εξήμιση λεπτά. Α, όχι, όχι, λέτε ψέματα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα την άποψή σας πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, διότι υπάρχουν δύο πτυχές του ζητήματος. Η μία λέει ότι όλες οι εργασίες πρέπει να είναι αξιοπρεπείς και η άλλη πλευρά λέει η εργασία είναι εργασία και πρέπει να τη δεχτεί κανείς. Ως προς το θέμα της ισότητας, το χάσμα διευρύνεται στα περισσότερα κράτη-μέλη. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εξάμεινο ως μέσο βελτίωσης. Η συνάδελφος από τη Δανία μίλησε για τη μη σωστή ανταπόκριση των ε, δεξιοτήτων. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν υπερβολικά προσόντα για μια θέση και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν αρκετά βεβαίως, αλλά υπάρχουν και αυτοί που διαθέτουν υπερβολικά πολλά προσόντα για μια θέση. Ο κύριος Λικιώτης ε, από την ΓΚΟΕ. Έχετε το λόγο. Ε, πρώτα απ' να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές ε, για τις ε, εισαγωγές τους ομιλίες. Ε, όμως πρέπει να αγγίξουμε τα προβλήματα στην ουσία τους και στη ρίζα τους με την έννοια ότι παρόλο είδα κριτικές απόψεις για αυτούς τους στόχους όσο συνεχίζονται οι πολιτικές της λιτότητας δεν μπορούμε να καλύψουμε τους στόχους. Ε, και σε ό,τι αφορά την ενεργεία και τη φτώχεια. Γιατί κακά τα ψέματα και δεν αναφέρομαι μόνο στις χώρες που πέρασαν από μνημόνια, αναφέρομαι σε όλα τα κρατημέλη, γιατί οι πολιτικές ζητότητας ε, δημιουργούν, ε, επιτείνουν την ύφεση, επιτείνουν την κρίση, καταργού θέσεις εργασίας. Είναι αλήθεια ότι αναφέρθηκαν οι ομιλητές και κυρίως η, κυρία Φρατσουάντε Μπόε για τα λίγα αποτελέσματα όσον αφορά την μείωση της φτώχειας και μάλιστα ε, φάνηκε ξεκάθαρα από την τοποθέτησή της ότι ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ε, για τα την άποψή μα, εμεί συμφωνούμε με του ομιλητέ που μίλησαν για την ανάγκη κοινωνικού διαλόγου και την άγκη να δουλέψουμε ε, συλλογικά στην κατεύθυνση τη καταπολέμηση τη φτώχεια, αυτό επαναλαμβάνω μπορεί να γίνει μόνο εάν οδηγηθούμε σε μια κοινωνική ανάπτυξη με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασία και βεβαίω ε, επειδή αναφέρθηκε και ε, η εκπρόσωπο από την ΑΛΤΕ, ε, ναι, για μα οι θέσει εργασία πρέπει να είναι αξιοπρεπεί και ασφαλεί. Η Ευρώπη έχει αυτή την ακατάκτηση, είναι κατάκτηση που έγινε με σκληρούς αγώνες εδώ και δεκαετίες και δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να οδηγήσουμε τους εργαζόμενους στην Ευρώπη στο επίπεδο των εργαζομένων που βλέπουμε στην περιφέρεια και στις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου ε, στο όνομα ότι πρέπει να γίνουμε ε, πιο ανταγωνιστικοί. Ε, γιατί τότε δεν θα εξυπηρετούμε καθόλου αυτό που θέλουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε κράτη δημοκρατικά, κράτη ευημερίας. Ε, είναι ανάγκη βεβαίω να αναθεωρηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, αλλά όπως είπα και προηγουμένως για να προωθηθούν ε, να προωθηθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσει εργασία, πρώτη θα πρέπει να γίνουν δημόσιε επενδύσει. Ε, το βλέπουμε σε πολλέ χώρε ότι οι ιδιώτε δεν ρισκάρουν. Θεωρούμε επίση λαθασμένο ότι γίνονται προσπάθειε να δημιουργηθούν κίνητρα για να επενδύσουν οι, οι μεγάλες ε, πολυεθνικές εταιρείες αλλά χωρίς να έχουν ρίσκο όπως το βλέπουμε και με το ε, πρόγραμμα, με το ε, πλάνο του κυρίου Γιούγκερ πριν να ολοκληρώσω θα ήθελα πρώτα πρώτα να, να ρωτήσω την άποψη των ομιλητών αναφερικά με τη σύνδεση, δηλαδή πώς βλέπουν τα ζητήματα της πολιτικής λιτότητας και των μνημονίων, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, ώστε να μην δημιουργούνται αποκλήσει από τους στόχους ε, για την απασχόληση και την εξάλληψη τη φτώχεια. Ήθελα δηλαδή τη δική του την άποψη. Το δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω την άποψη του κυρίου Βάιζε αναφορικά με το ντάμπινγκ μισθών που παρατηρείται στη Γερμανία και πω αυτόν επηρεάζει την απόκληση από του στόχου για την απασχόληση και την εξάλληψη τη φτώχεια στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το, στον κύριο Μάρτε. Ε, προσπαθήσατε να μας αποκρύψετε ότι έχετε γενέθλια, αλλά εμείς ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. And then I'll give the floor to Laura Agia from EFTD Group. Grazie Presidente, e grazie. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ομιλητές που μας έδωσαν μία συνολική εικόνα, μία εγκάρσια εικόνα που σχετίζεται με διάφορες πτυχές της στρατηγικής. Είδαμε και τις διάφορες προοπτικές που διανοίγονται. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις και ίσως μπορούμε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο. Καταρχήν, στην εκπρόσωπο των Σουηδικών Συνδικάτων θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση μεταξύ πολιτικής και συνδικάτων στη χώρα της, γιατί είναι σαν να μου ανοίχτηκε ένας κόσμος ο οποίος είναι άγνωστος για τη χώρα μου. Και γι' Το πιστεύω ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι δεν εισακούνται μόνο ε, κατακαιρματισμένα, αλλά εισακούνται γενικότερα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη χώρα μου. Στη χώρα μου τα συνδικάτα είναι οι προμαχώνες των πολιτικών κομμάτων. Αρχίζει κανείς από συνδικαλιστής και στο τέλος γίνεται πολιτικός, επαγγελματίας πολιτικός. Ποια είναι η οριοθέτηση λοιπόν σε εσά όσον αφορά την σουηδική διάσταση. Στη συνέχεια άκουσα για μη τυποποιημένη εργασία, για άτυπη εργασία Δηλαδή ας αρχίσουμε να εργαζόμαστε ε, χάρη της εργασίας και μόνο. Εγώ είμαι της γνώμης ότι ε, αν μειοδοτήσουμε ως προς αυτή την ε, αρχή, τότε ο κανόνας αυτός θα παγιωθεί. Και ε, αν αρχίζουμε με αγαθές προθέσεις, Στη συνέχεια θα ε, μεταφερθεί, θα γίνει μάλλον αυτή η εργασία ένα καρκίνωμα από το οποίο δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε. Όταν μιλάμε για εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούνται σε αυτά τα φόρα όταν οι πολίτες ε, γίνονται μέλη των θεσμικών οργάνων, όταν δεν ξεχνούν ποιοι είναι και από πού προέρχονται. Έγινε λόγος για τους ε, δείκτες απόλυτης ε, φτώχειας ως μία μορφή αποκλεισμού του κινδύνου, ε, κοινωνικού αποκλεισμού, απόλυτου κοινωνικού αποκλεισμού. Αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για κοινωνικούς δείκτες φτώχειας, τι μας προτείνετε, τι μας υποδεικνύεται για να ορίσουμε σαφή στοιχεία. Γιατί ειλικρινά εδώ και ένα χρόνο η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα αφορά τον ορισμό κοινωνικών δικτών για τη φτώχεια, για την οριοθέτηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε λόγος και για εξάντες συντονισμό των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να δούμε ποιες θα είναι η... ποια θα είναι η αποδοτικότητά τους. Ναι, αυτό έπρεπε να γίνει εξ αρχής. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση εξάντε. Μπορεί μόνο να γίνει μια εξπόστα αποτίμηση. Γιατί η κοινωνική σφαγή ε, βρίσκεται υπό το βλέμμα όλων μας. Ίσως μερικά χρόνια πριν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτή την εξάντε αποτίμηση, μια πολιτική πρόληψη δηλαδή. Σήμερα μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, ε, άκουσα και κάτι άλλο, αλλά σποραδικά Ένας από τους στόχους του εξαμήνου είναι να επιλύσουμε τη μακροχρόνια ανεργία, γιατί από εκεί απορρέει σωρία προβλημάτων. Η παιδική φτώχεια είναι απότοκη της ε, μακροχρόνιας ανεργίας. Γονείς που δεν εργάζονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να εγγυηθούν την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών. Ποιες είναι οι υποδείξεις ε, ως προς αυτή την πτυχή του θέματος, έπειτα ως προς το ανθρώπινο μυαλό. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την παρέμβαση του καθηγητή Καπέλο, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στη χώρα μου και θα τελειώσω με αυτό. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε να κάνουμε με πραγματικότητες που χρησιμοποιούν αυτές τις καινοτόμες ιδέες. Δηλαδή η χαρτογράφηση του νου χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια καινοτόμων σχεδίων για να δοθούν αποτελεσματικές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα σε δύο μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Γουαρνταρούμπια Ζαμπάλ. από τους σοσιαλδημοκράτες, την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών επίσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι είμαι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και γι' αυτό θα ήθελα να θέσω στους συζητητές ε, κάποιες ερωτήσεις. Πώς βλέπουν δηλαδή την σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 2020 και την αντιστήχησή τους με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τα προβλήματα έλλειψης, ελλείψεων δημοσιονομικών ε, ιδιαίτερα για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες για το πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020 με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς στην φάση αυτή θα κάνει, ετοιμάζει μάλλον κάποιες προτάσεις για τα δημοσιονομικά για τα επόμενα χρόνια, για την παρούσα δημοσιονομική περίοδο και θα ήθελα να μάθω με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, μέσω ποιων προγραμμάτων θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Thank you. Uh, uh, Ο κύριος Μαραγκάλ από πλευράς των Πρασίνων. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς μιλάμε περισσότερο για τα αποτελέσματα και όχι τόσο για τις αιτίε. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, νομίζω ότι στην ουσία φτάνει αυτό. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς λόγους που δημιουργούν ανισότητες, που δημιουργούν ακραία φτώχεια και ανεργία. Και αυτό επηρεάζει με δραματικό τρόπο την ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων Ακούσαμε εξαιρετικές παρεμβάσεις από χώρες όπως η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, αλλά να σκεφτούμε λίγο τι μπορεί να συμβαίνει και σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ουσία η πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταποκριθούν και στη συνέχεια ε, δείχνουμε ότι εκπλησόμεθα όταν υπάρχει μείωση δημοσίων υπηρεσιών. Μετά προσφεύγουμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προβάλλουμε κυρώσεις στα κράτη-μέλη τα οποία δεν προβάλλουν τα σωστά πλαίσια κυρώσεων. Μετά μιλάμε για το σχέδιο Juncker όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε την, ε, τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εισαγάγει ούτε ένα ευρώ στον προϋπολογισμό της. Πρόκειται για ένα σχέδιο χωρίς ε, περιφερειακές ποσοστώσεις αλλά και χωρίς εξισορροπημένη στρατηγική. Ε, μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία. Φυσικά αυτό μας ενδιαφέρει. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους σωστούς όρους για να αντιμετωπίσουμε την συγκεκριμένη ενδοκινοτική μετανάστευση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους εισηγητές ε, κατά πόσο δέχονται τις ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και κατά πόσο θα πρέπει να προβάλλουμε τις ε, διάφορες ανισότητες οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Δεν θα έπρεπε να προβάλλουμε μία σωστή πολιτική για την αντιμετώπιση της ε, διαρθρωτικής ανεργίας. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μία ε, πρόκληση που σχετίζεται όχι μόνο με την αναθεώρηση της στρατηγικής, αλλά και με την διάθεση μιας πραγματικής μεταρρύθμισης εις βάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τεμπόου είπε στην εισαγωγή της ότι οι επιπτώσεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι αμεληταία Τώρα υπάρχει σωρία ερωτήσεων με το ίδιο θέμα και μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως μπορείτε να απαντήσετε. Αρχίζουμε με τον κύριο Βάισε. Ξέρω ότι είναι αδύνατον να είσαστε σύντομοι, αλλά θα ήθελα να το προσπαθήσετε με θέματα μίζωνος σημασίας και να είσαστε ιδιαίτερα λακωνικοί. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις και θέσεις σχετικά με το ποιες είναι οι τυπικές θέσεις εργασίας. Έχουμε τις επισφαλείς ε, ε, θέσεις εργασίας και υπάρχει μια αναγνώριση ότι διάφορες μορφές μερικής απασχόλησης έχουν ε, μειώσει την ανεργία, έχουν αυξήσει την απασχόληση. Ωστόσο, από αυτήν την είσοδο στις αγοράς εργασίας ε, δεν ε, βλέπουμε ε, σαφή άνοδο εντός της αγοράς εργασίας. Δεύτερον, οι τυπικές και άτυπες θέσεις εργασίας δεν θα ισχύουν στο μέλλον. Σήμερα στο ίντερνετ έχουμε μορφές εργασίας όπου κάποιος ε, κάνει login, συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα, πληρώνεται χωρίς συνεισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φορολογία κλπ. Οι τυπικές και άτυπες θέσεις δηλαδή είναι όροι που δεν θα καλύψουν τις μορφές αυτές στο μέλλον. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που απέναντι στους πολίτες τους δεν προσφέρουν ε, ελάχιστο επίπεδο όπως άλλα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, καθόλου επαγγελματικό προσανατολισμό στο σχολείο. Η βοήθεια με στόχο την αυτοβοήθεια ή την συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και απασχολούμενων όσον αφορά την απασχόληση που στοιχίζει ε, για όλους. Ε, είναι κάτι όμως που επίσης προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον. Επίσης όσον αφορά την απασχόληση θα πρέπει να πούμε ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι ευέλικτος όσον αφορά την επιλογή της απασχόλησης να είναι κινητικός και να ενδιαφέρεται για μετεκπαίδευση. Χωρίς αυτά δεν θα πετύχουμε αυτό που, επιθυμούν, που επιθυμούμε. Όσον αφορά την πολιτική λιτότητας, Μπορώ να μιλήσω μόνο εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης της Γερμανίας και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρχαν λοιπόν επί χρόνια σημαντικά ελλείμματα. Με τα χρόνια μάθαμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να επενδύουμε μόνο εκεί όπου έχουμε αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν έχουμε επαρκείς πόρους για τους νέους, επαρκείς δομές και πολλά μέρη όπου μπορούμε να στηρίξουμε νέους ανθρώπους. Μέσα σε 10 χρόνια καταφέραμε να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας των νέων. Αυτό το πετύχαμε με τις σωστές δομές και κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαμε ελάχιστες επιπτώσεις, διότι είχαμε τις συνεισφορές εργοδοτών και εργαζομένων με τις οποίες μπορέσαμε να στηρίξουμε τον κόσμο ώστε να μην γίνουν τόσες απολύσεις. Βλέπω λοιπόν ότι πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν τέτοιες δομές. Δεν αξίζει τον κόπο να επενδύουμε πολλά χρήματα σε κακές δομές τα δύο τρίτα της μακροπρόθεσμης ανεργίας στην Γερμανία χαρακτηρίζεται από ανθρώπους που δεν έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα και είναι άνω των 50 ετών. Εγκαίρως λοιπόν να φροντίσουμε να έχει ο κόσμος επαρκή εκπαίδευση. Αδυναμία στη Γερμανία αποτελεί το ότι υπάρχει ακόμα προκατάληψη όσον αφορά τους πιο ηλικιωμένους. Είμαστε ευγνώμονες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετά την επανένωση της Γερμανίας απορρόφησαν χιλιάδες νέων από την προενατολική Γερμανία και τους, και τους προσέφεραν θέσεις εργασίας. Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό είναι πολύ ε, θετικό μήνυμα για την Ευρώπη. Πολλοί κόσμος δεν ξεχνά την πατρίδα του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τεμπόη. Ευχαριστώ. Για τα θέματα της απασχόλησης με τις ερωτήσεις που μου κάνετε, πράγματι ποιοτικέ θέσει απασχόλησης, αυτό επιδιώκουμε. Θέλουμε όμως να στοχεύσουμε και σε ένα επίπεδο όχι αυστηρά μακροοικονομικό. θα μπορέσουμε ίσως να μπούμε σε μια τέτοια λογική αφού εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε σωστά τους εργαζομένους για να μπορούν να βρουν κάποια θέση ικανοποιητική. Αυτό μπορεί να καλύψει και την κατηγορία των λεγόμενων μη τυπικών θέσεων εργασίας για τα θέματα της λιτότητας. Στο Βέλγιο είμαστε μια χώρα που την έχει λίγο γλιτώσει μέχρι τώρα αυτό έγινε χάρη στην κοινωνική προστασία που έχουμε και που μας έχει προστατεύσει από τα φαινόμενα της κρίσης που είχαμε εν μέρη και εδώ. Αλλά η τάση είναι μείωση ε, των ρυθμίσεων προστασίας και για τη μείωση των επιδοτήσεων για την ανεργία και της διάρκειας ε, χορήγησης των επιδομάτων αυτών και υπάρχουν ε, και πραγματικά μια κατηγορία ανθρώπων, υπάρχουν άνθρωποι που χάνονται από όλα τα δίκτυα προστασίας. Περνούν από κάποια δίκτυα και κάποια στιγμή τα δίκτυα τους πετάνε έξω και εξαφανίζονται. Οπότε εκεί δεν τίθεται πλέον θέμα προστασίας. Τώρα για την συμματοχή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό. Εμείς στη δική μας υπηρεσία προσπαθούμε να, να προετοιμάζουμε τις συναντήσεις αυτές. Είναι δύσκολο να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς που είναι εκτός εργασίας να έλθουν σε επαφή μαζί μας, να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους και δεν μπορούμε να κάνουμε την σωστή προετοιμασία που θέλαμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζουν με στη φτώχεια έχουν τις γνώσεις που θα ήταν χρήσιμες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι απόλυτα διατεθειμένοι να συμμετέχουν. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε τους τρόπους συμμετοχής και έτσι κι αλλιώς μία μεγάλη συνάντηση το χρόνο φυσικά δεν αρκεί από μόνη της. Νομίζω ότι απαιτούνται πιο τακτικές συναντήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς υπευθύνους, στους υπαλλήλους και στους, στις, στους συλλόγους που ασχολούνται με τα θέματα φτώχειας. Ευχαριστώ κυρία Νίγκρεν. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στην συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με την σχέση ανάμεσα στις καλλιστικές οργανώσεις και την πολιτική στη Σουηδία. Όπως είπα και στην παρουσίασή μου, έχουμε τρεις κεντρικές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες στην ε, Σουηδία. Και σε αντίθεση με πολλά άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η οργάνωση γίνεται όχι ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση, αλλά με τον τομέα στον οποίο εργάζονται τα μέλη μας. Ε, φυσικά προσπαθούμε να επηρεάσουμε την πολιτική, αλλά κυρίως διαπραγματευόμαστε όσον αφορά την σχέση με τους εργοδότες. να περάσω στι γενικέ ερωτήσει που συστήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια τη ακρόαση. Θα ήθελα να συνοψίσω το μήνυμά μα ω εξή. Οι στόχοι τη στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι καλοί, δεν είναι επαρκή όμω. Συμβουλή προς τους πολιτικούς. Θα πρέπει να έχουμε σωστές επενδύσεις, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την ζήτηση, την οικονομία και να έχουμε μια πολιτική που να προωθεί τα θέματα αυτά. Η και πολιτική προς όφελος των ανθρώπων. Η κοινωνική ασφάλεια δημιουργεί ε, παραγωγικότητα, ένα σύστημα όπου ε, να νιώθει κανείς ασφαλής, όπου να μην εργάζεται ε, αν για παράδειγμα είναι άρρωστος. Θα πρέπει να μπορεί κανείς να αγοράζει τα τρόφιμά του, να πληρώνει τον νίκη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπως και η μισθή. Η φτώχεια συνδέεται με το θέμα των ε, θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Χρειάζονται θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. Σε όλη την Ευρώπη τον τελευταίο καιρό αυξάνεται η φτώχεια εργαζομένων, δηλαδή πολύ χαμηλός μισθός ώστε να μην μπορεί κανείς ε, να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του. Και μάλιστα συμβάσεις εργασίας ε, με ελάχιστες ή και μηδενικές ώρες εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προωθήσουμε την παραγωγικότητα και την οικονομία. Κλείνοντας, η σημαντική στόχη τη στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλε τι πολιτικέ, ώστε η κοινωνική πολιτική ή η πολιτική απασχόληση να μην είναι απλά διακοσμητικά, ώστε να μπορούμε να περάσουμε στο κοινό πολιτικέ που δεν είναι προ όφελό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέλφερη, έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον που δίδεται βάση στα θέματα της πολιτικής απασχόλησης. Και ξανά στρέφουμε την προσοχή μας στα συστήματα κοινωνικής προστασίας που έχουν ε, υποφέρει από την κρίση και που μπορεί να βοηθήσουν έτσι ώστε να δοθεί εκ νέου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που λείπει μερικές φορές σε αυτούς οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από την ε, οικονομική κατάσταση. Η δυσκολία είναι πολλές φορές την είσοδο στην ε, αγορά εργασίας. Ε, η απασχόληση βέβαια από μόνη της κάτω από συγκεκριμένες μορφές δεν είναι πανάκια, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να υπάρξει μια θέση εργασίας η οποία να ικανοποιεί και να καλύπτει τις ανάγκες. γιατί ξέρετε ότι όσο είναι κάποιος εκτός εργασίας, όσο περνά ο καιρός μειώνονται οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις και όλο και περισσότερο ε, βυθίζεται κανείς σε μια θάλασσα από χρέος και απογοήτευση. Συνεπώς λοιπόν ε, πρέπει να υπάρξει σωστή προετοιμασία για τους ανθρώπους αυτούς που θα ξαναβρούν μια κάποια θέση απασχόληση. Τώρα οι μεταρρυθμίσεις έτσι όπως προτείνονται έχουν σαν μοναδικό στόχο την ανταγωνιστικότητα και αυτό φυσικά πιέζει α, ε, τις αμοιβέ, τους μισθούς, αυξάνει βέβαια την κινητικότητα των εργαζομένων αυξάνει αυτούς οι οποίοι δουλεύουν αλλά είναι φτωχοί και αυξάνει και τον αριθμό αυτών που έχουν δύο θέσεις, δύο α, μορφές απασχόλησης. Ένα άλλο θέμα είναι να δούμε και τι γίνεται με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των συντάξεων, να δούμε τι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στους πολίτες και ιδιαίτερα στις γυναίκες αν περάσουμε από το ένα σύστημα στο άλλο, κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις εξελίξεις. Άκουσα με ενδιαφέρον βέβαια επανειλημμένα ότι απαιτείται να υπάρξουν μελέτες επιπτώσεων για το τι κάνουν οι μακροοικονομικές πολιτικές, στις κοινωνικές πολιτικές σήμερα ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ήδη ζουν με στη φτώχεια ή σε κίνδυνο φτώχειας. Είναι κρίσιμο να υπάρξει μια ετήσια έκθεση η οποία να παρακολουθεί όχι μόνο την εφαρμογή αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις ετήσιες αναχώρα συστάσεις και πώς έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις αυτές για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, για την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της ήταν μια απογοήτευση. Στην αρχή χαιρετίστηκε σαν μια διαδικασία, όχι σαν ένα συμβάν σε αιτήσια βάση, αλλά σαν μια διαδικασία για παρακολούθηση των στόχων της φτώχειας. Αυτό δεν συνέβη δυστυχώς και τώρα περιμένουμε νέες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να οργανώσουμε με διαφορετικό τρόπο τον διάλογο αυτό, ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν προβλήματα φτώχεια σήμερα. Συναντώνται βέβαια άπαξ σε αιτήσια βάση αλλά η διαδικασία δυστυχώς έχει πάρα πολλά κενά και πρέπει να επανεξεταστεί έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορέσει να μπει σε διάλογο με τους θεσμούς και να ευημερήσουν όχι μόνο οι αριθμοί αλλά και οι πολίτες οι οποίοι φύγονται σε εθνικό επίπεδο. Για τους πίνακες αποτελεσμάτων φυσικά πάντα θέλαμε να υπάρχει ένα τέτοιο scoreboard και ένα μηχανισμό ε, νομικό για διορθωτικές δράσεις. Και τέλος η, η ε, ενδιαφέρουσα ερώτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε για τα θέματα χρηματοδότησης. Εμείς θέλουμε να συνδυάσουμε το κοινωνικό ταμείο ε, και προγράμματα όπως το Horizon για να στηρίξουμε τις κοινωνικές πολιτικές και να δώσουμε περισσότερους πόρους στην κοινωνία των πολιτών και στις οργανώσεις της που βοηθούν στην εφαρμογή και επίτευξη αυτών των στόχων. Λοιπόν, τρία δις για το Ταμείο Εγγυήσεων για τον Νέο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη γύρω από αυτό και δεν έχουμε στοιχεία για χώρες από τις μεμονωμένες εκθέσεις γύρω από το Ταμείο των Νέων. Ευχαριστώ. Καπέλο. Ευχαριστώ. Τα θέματα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να πω ότι είναι και ιδιαίτερα δελεαστικά. Αρχίζουμε από το θέμα της απασχόλησης. Δεν ξέρω την ε, κατάσταση σε άλλες χώρες, αλλά ξέρω την κατάσταση στην Ιταλία, τη χώρα μου. Η άτυπη εργασία ξεκίνησε σαν ε, μία δυνατότητα, να, μία ευκαιρία να μπει κανείς στο χώρο εργασίας. Έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς ε, δεν εξελίχθηκε έτσι. Αυτό οδήγησε σε έλλειψη εμπιστοσύνης του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων. Όσο αφορά τη λιτότητα, ε, ζητήσατε τις σκέψεις μας, τις σκέψεις του πάνελ. Εγώ είδα να ε, πλήττεται ιδιαίτερα το σχολείο, τα σχολεία, η εκπαίδευση. Και φυσικά αυτό ε, στην ουσία έπληξε την κατάρτιση και την εκπαίδευση ως ευκαιρία δημιουργίας θέσεων εργασίας σε σχέση με την ε, απόσταση μεταξύ στόχων και απολογισμού. Όπως είπε και ο Ευρωβουλευτής από την Επιτροπή προϋπολογισμών μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι δεν έχει σημασία μόνο να δαπανούμε χρήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι από πού θα αντλήσουμε τα χρήματα και πώς μπορούμε να καταρτήσουμε τους ανθρώπους, να προβούμε σε έναν αλφαβητισμό έτσι ώστε να ε, δημιουργηθεί ένας μοχλός να χρησιμοποιηθεί μάλλον αυτός ο μηχανισμός ως μοχλός. Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας και αυτό έχει να κάνει και με μία διαδικασία απλούστευσης. Αυτό ε, έχει σχέση και με την εμπιστοσύνη των πολιτών. Προτείναμε λοιπόν προτείναμε να υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια. Το Cambridge και η Oxford προτείνουν τέτοια σχήματα και αυτό αφορά και πανεπιστήμια των ΗΠΑ και καναδικά ε, πανεπιστήμια που προτείνουν προγράμματα ε, ε, map minding. Ο δόκτωρ Νίκη Όπενχάιμερ είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Είναι ο πρόεδρος της Debers, ενός μεγάλου ε, κολοσσού παγκοσμίως. Επίσης, το Υπουργείο Εξοπλισμών της Νέας Ζηλανδίας που χρησιμοποιεί αυτές τις ε, τεχνικές mind mapping. και ο Μπέντζαμιν ε, Τζάντερ που είναι ο διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βοστόνης, όλοι αυτοί οι τομείς, δηλαδή οι τομείς που καλύπτουν ένα ευρύ ε, γνωσιακό φάσμα, δημιουργούν αυτές τις, χρησιμοποιούν αυτές τις ε, τεχνικές και αυτό μας ανοίγει και τους ορίζοντες ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσεν από τη Δανία. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω τις ερωτήσεις σε τρεις-τέσσερις ομάδες. Καταρχάς, όσον αφορά την απασχόληση. Μιλώ ως Δανέζα. Στη Δανία έχουμε το μοντέλο της ελαστασφάλειας, το flexibility. Έχουμε μια ανοιχτή και δυναμική αγορά εργασίας, όπου ο κόσμος τολμά να αλλάξει δουλειά. στη Δανία. Έχουμε 800.000 ε, ε, ε, ευκαιρίες απασχόλησης το χρόνο, που είναι πάρα πολύ για μια χώρα με 5 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο από τις θέσεις που καλύπτονται κάθε μέρα καλύπτονται από ανέργους. λέξη κλειδί είναι η ανοιχτή και δυναμική αγορά εργασίας, ώστε ο κόσμος να τολμά να αλλάξει θέση, να βρει μια καλύτερη δουλειά με περισσότερες ευθύνες, περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερη αμοιβή κλπ. Νομίζω ότι από τους φιλελεύθερους τέθηκε ερώτηση σχετικά με το ότι σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε ανθρώπους με υπερβολικά προσόντα σε σχέση με την θέση απασχόλησής τους. Δηλαδή έχουν πάρα πολλές δεξιότητες, ε, αλλά δεν βρίσκουν ε, αντίστοιχη θέση εργασίας. Πιστεύω ότι το benchmarking μπορεί να αποτρέψει τέτοιες καταστάσεις και νομίζω ότι έχουν υπάρξει τάσεις σχετικά με τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σχετικά με το 40%. Νομίζω ότι επικεντρωθήκαμε πολύ περισσότερο στις, ε, στην ανώτερη εκπαίδευση, διότι υποτίθεται ότι έχει πιο πολύ πρεστής μια, μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση από επαγγελματική κατάρτιση. Μία δυνατότητα θα ήταν να δημιουργήσουμε μία τριμερή συνεργασία ώστε οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις, η κυβέρνηση ε, να συνεργάζονται και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να σκεφτούν τι χρειαζόμαστε στο μέλλον. Διότι είναι απαραίτητο να γίνεται με αυτόν τον τρόπο τελευταία ομάδα ερωτήσεων στην οποία θα ήθελα να απαντήσω έχει να κάνει με τους μηχανισμούς κινητοποίησης ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν και να εφαρμόζουν τις συστάσεις αναχώρα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με πιο επικοδομητική χρήση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουμε κίνητρα και ποινές. όταν για παράδειγμα μια χώρα εφαρμόζει τις ε, συστάσεις αναχώρα να λαμβάνει ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να συνδέσουμε την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ξέρει ότι έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα ε, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαγγελματική κατάρτιση, για παράδειγμα, ε, ενώ οι χώρες δεν έχουν ζητήσει τα χρήματα αυτά. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές, στους οποίους θα δώσω το λόγο τώρα. Την κυρία Σαντέρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την κοινωνική κατάσταση στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κατάσταση η οποία μας παρουσιάστηκε σήμερα. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε μια νέα έκθεση στη Γαλλία, στη χώρα μου, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση πραγματικά φτώχειας και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι η κατάσταση, όπως είπαν κάποιοι ήδη, περνά μέσα από την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και δίδοντας πρόσβαση στην απασχόληση, τότε μόνο θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την φτώχεια γιατί η απασχόληση φυσικά δίδει εισόδημα αλλά ταυτόχρονα δίνει και αξιοπρέπεια. Μια κατοικία, μια στέγη δίνει επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικές όπως υπηρεσίες υγείας κτλ. Η πρόσβαση στην απασχόληση θα επιτρέψει να ρυθμιστούν κάποια από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα επιτρέψει επίσης να προχωρήσουμε ε, πετυχαίνοντας τους στόχους της Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Η κατάσταση σήμερα χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορροπίας στο εσωτερικό της Ένωσης. Υπάρχουν ορισμένες χώρες μέλη με ιδιαίτερα υψηλή ανεργία και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Έχουν προταθεί διαφορετικές λύσεις δεν νομίζω ότι υπάρχει μία μόνη λύση. Εγώ θα ήθελα να προτείνω κάποιες, αλλά ξέρω ότι πολλές από αυτές έχουν ήδη τεθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι απαιτείται μία λύση εν μέρη ευρωπαϊκή, εν μέρη εθνική. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή λύση θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο όπως ε, υπόθηκε ήδη από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτείται να υπάρξει μια καλύτερη λήψη υπόψη των κοινωνικών δικτών. Οι κοινωνικοί δείκτες είναι αυτοί που θα μας ε, δώσουν την εικόνα των κρατών μελών. Το θέμα το οποίο τίθεται είναι αν οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να καταστούν δεσμευτικοί, γνωρίζοντας ότι σήμερα Κάποια από αυτά τα κοινωνικά θέματα δεν ανήκουν σε κοινοτικές αρμοδιότητες, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι δεσμευτικοί μακροοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι όμως δεν γίνονται σεβαστοί από τα κράτη-μέλη. Οπότε τι είδους δεσμευτικοί είναι αυτοί οι κανόνες. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν για τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις ειδικέ αυτές ρυθμίσεις χώρα και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ανάγκη να ρευστοποιήσουμε κάπως περισσότερο την αγορά εργασίας και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο πιέζοντας τα κράτη-μέλη. Μία τελευταία λέξη πρόεδρε. Να πω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο για τοπικές λύσεις για να ευνοήσουμε ακριβώς ε, την κατάρτιση, την μαθητεία και να μην αγνοούμε ε, μέτρα τα οποία μπορεί να ληφθούν σε επίπεδο ε, συνοριακό μεθοριακό. Κύριος Μαρτάν έχει το λόγο. Και εγώ ονομάζομαι Μαρτάν, αλλά Εντουάρ. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί ε, μου ευχηθήκατε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την βεβαιότητα μερικών που χρησιμοποίησαν ε, στερεότυπα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν χώρες που κράτησαν ε, αυτούς ε, τους ε, κοινωνικούς σταθμιστές και άλλες που χρησιμοποίησαν την απορρίθμιση που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει σιγουριά για το τι λειτουργεί και τι όχι. Επίσης άκουσα και κάτι άλλο από όλους τους παρεμβαίνοντες. Μα τι θα πει ποιοτική εργασία. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ποιοτικό μισθό. Δεν υπάρχει κανένας αυτόματος συσχετισμός μεταξύ ε, εργασίας ε, και απομάκρυνσης από τη φτώχεια. Ξέρουμε πολλούς φτωχούς ε, μισθωτούς που δεν έχουν ούτε καν στέγη, άρα δεν υπάρχει συσχετισμός. Ας μιλήσουμε για ποιοτικούς μισθούς και έναν ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό που να καλύπτει όλους, γιατί θα πρέπει να δούμε τι θεωρείται ποιοτική εργασία. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένες εργασίες που ε, δεν τις θέλει ο κόσμος γιατί έχουν άτυπα ωράρια. Στη Γαλλία γνωρίζουμε ανάπτυξη αλλά χωρίς εργασία. Βεβαίως υπάρχει παραγωγικότητα και επενδύσεις οι οποίες είναι περιορισμένες όμως. Υπάρχει ε, χρόνια έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και τα, το έλλειμμά μας και το χρέος και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια, ποιοι είναι οι φτωχοί συγγενείς. Δηλαδή η καταπολέμηση της ανεργίας είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και το κόστος εργασίας. Εάν ε, στην Ισπανία υπάρχουν, περικές, ε, ε, περι, υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, αυτό έγινε γιατί μειώθηκαν οι μισθοί σε αυτό τον φαύλο ε, κύκλο δεν υπάρχει λύση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντερό το εξής. Μιλήσατε για την ε, κοινωνική ρήτρα, την οριζόντια κοινωνική ρήτρα και για την καταπολέμηση της φτώχειας, πώς μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε καλύτερα αυτό το μέσο για να είναι πιο αποδοτικό. Τέλος, η τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Μαν. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Βάιζε, θα ήθελα να επικεντρωθώ στη δική σας παρέμβαση. Σπάνια. Στο Κοινοβούλιο ακούμε γιατί πότε πότε είναι καλό να εξοικονομεί κανείς χρήματα. Ε, μιλήσατε για την αποτελεσματική επένδυση των χρημάτων. Σημαντικό είναι να κάνουμε οικονομίες ώστε να μπορούμε να τα επενδύσουμε την κατάλληλη στιγμή. Και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εκλογές ε, όπου το αποτέλεσμα είναι ε, εξτρεμιστικό είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Αυτό είναι τελείως λάθος. Στην πολιτική θα πρέπει να πούμε σταματήστε την πολιτική λιτότητας. και υποσχεθούμε στους πολίτες ένα σωρό πράγματα. Αυτό είναι πολύ καλό για αυτούς που σκέφτονται μόνο τις εκλογές, αλλά θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε στο ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι καλό πότε πότε να έχουμε και μία περίοδο λιτότητας ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε αποτελεσματικά τα χρήματα την κατάλληλη στιγμή. Και ο κύριος ε, Καπέλο, ε, είπε, μίλησε πολύ σωστά. Το θέμα δεν είναι είτε λιτότητα είτε επενδύσεις. Τα πράγματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και πολύ σωστά είπε ο Ζων Κλοντ Ιούνκερ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα των 350 δισεκατομμυρίων διότι εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα, εκεί θα πρέπει να γίνονται οι επενδύσεις, όχι όμως να πετάμε τα χρήματα με τον κουβά. Πολλοί διεθνείς ε, φορείς, πολλοί διεθνείς φορείς ε, έχουν τις ε, ίδιες αρχές, αλλά στην Γερμανία τι βλέπουμε. Βλέπουμε μεγάλη ανεργία για τους άνω των 50. Βλέπουμε όμως και διαρροή εγκεφάλων, ψυλές γνώσεις, Έχουμε σημαντικές απώλειες στους νέους μας. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν να προοδεύσουμε, γιατί δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να πούν ότι θα προσλάβω ανθρώπους πιο ηλικιωμένους διότι είναι αξιόπιστοι ε, και δεν θα μου φύγουν ε, αύριο. Γιατί λοιπόν δεν προχωράμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς την κυρία Ντεπόε ακούσαμε ε, και οι υπόλοιποι θα αποφασίσετε εσείς οι ίδιοι αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που ακούσαμε. Κυρία Ντεπόε παρακαλώ. Ευχαριστώ σε σχέση με το οριζόντιο κοινωνικό, με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι η επίπτωση του κανονισμού για τη φτώχεια. Εγώ δεν δουλεύω στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ξέρω ότι δεν λειτουργεί πολύ καλά. Μπορώ να σας πω τι συμβαίνει στο Βέλγιο το Ομοσπονδιακό κράτος έχει έναν κεντρικό κανονισμό και μετά οι περιφέρειες βλέπουν πώς θα τον εντάξουν και βλέπουμε σε ομοσπονδιακό επίπεδο ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να δίνεται νέα όθηση συνέχεια γιατί κάθε φορά που προβλέπεται ένα μέτρο εξάντε ζητάμε από τους υπαλλήλου να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις επιπτώσεις για την ε, φτώχεια. Αλλά οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ε, το θέμα της φτώχειας, γι' αυτό θα πρέπει να επινοήσουν την απάντηση αν και δεν έχουν τα μέσα. Ένα από τα ζητήματα που συζητάμε τώρα είναι η κατάρτιση, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση για την επίπτωση, της επιπτώσεις της φτώχειας, όπου να γίνονται και συζητήσεις, γιατί αν θέλουμε να γνωρίσουμε την ουσία της διαδικασίας που δεν αφορά μόνο τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, θα πρέπει να υπάρχουν και ποιοτικέ δοκιμασίες και θα πρέπει να πω ότι στο Βέλγιο υπάρχει διαφάνεια, τα, τις δοκιμασίες αντικτύπου τις βλέπει ο καθένας στο διαδίκτυο, αλλά δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος, υπάρχει μόνο ή θετικός ή ουδέτερος. Θα πρέπει λοιπόν οι υπάλληλοι να μπορούν να έχουν ποσοτικά στοιχεία που να τα μετατρέψουν σε ποιοτικά. Και επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε, να δώσουμε χρόνο έτσι ώστε να γίνει μία επισκόπηση επιτόπου. Είναι κάτι το ιδιαίτερα περίπλοκο, θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα μέτρα ε, παρά να συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια. Δεν ξέρω τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω μάθει ότι δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτό το πλαίσιο. Ίσως θα πρέπει να τύχει βελτίωση. Ο κύριος Βάης. Ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με, τις, με τα αρνητικά φαινόμενα, τους ε, χαμηλούς ε, μισθούς ε, και τις κακής ποιότητας θέσης εργασίας. Ένα κλειδί υπάρχει πάντα, να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Αυτό συνδέεται με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ψηφιοποίηση, έχει να κάνει με το πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει Ε, το εργατικό δυναμικό και στηρίζει τους απασχολούμενους. Σε πολλές χώρες έχουν γίνει διαπραγματεύσεις από τους κοινωνικούς εταίρους, από τις επιχειρήσεις δηλαδή και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που στο κάτω-κάτω καλύτερα από όλους γνωρίζουν ε, ε, την αξία των πραγμάτων. Στην Ευρώπη δεν είναι ο στόχος μας η λιτότητα. Στόχος είναι να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, δηλαδή με τα χρήματα που επενδύουμε να πετύχουμε στόχους, να δημιουργήσουμε καλύτερες δομές. Η οικονομία είναι πάντα να συγκρίνουμε τις διάφορες λύσεις για να βρούμε την καλύτερη σοκάρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει πόρους για τα ελάχιστα πρότυπα της εγγύησης για την νεολαία. Πολλές χώρες όμως δεν έχουν υποβάλει αίτηση για να ζητήσουν τα χρήματα αυτά, να διακριτήσουν τα χρήματα αυτά. Οι συνάδελφοί μου λοιπόν θα πρέπει να κάνουν το βήμα αυτό για την εφαρμογή των προγραμμάτων, διότι οι πολίτες δεν πρόκειται να δεχτούν τίποτα άλλο. Θα πρέπει επίσης να προβλέπουμε ευέλικτη απόσυρση από την αγορά εργασίας ε, και όχι διακοπή. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τις ηλικιωμένου και θαυμάζω τις χώρες που παρέχουν τέτοιου είδους ευελιξία. Μπορεί στη Γερμανία να μην τα κάνουμε όλα καλά, θα πρέπει να εξετάσουμε όμως τι κάνουμε σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ευέλικτες δομές. εργαζόμαστε όλο και περισσότερα χρόνια, αλλά κάποιος που γίνεται άνεργος στα 59 του δεν έχει πολλές ευκαιρίες να επανέλθει στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για σας. Σας ακούσαμε με ενδιαφέρον. Είμαστε η Επιτροπή Απασχόλησης και Θέματα Κοινωνικά. Έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά τα οποία για μας είναι πολύ όπως είπα σημαντικά. Ακούσαμε και είδαμε μάλλον ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χρήσιμες παρατηρήσεις. Σημείωσα 18 θέματα επιμέρους. Δεν είναι εύκολο για μας που εργαζόμαστε με τα θέματα αυτά σε πολιτικό επίπεδο αλλά νομίζω ότι η κατάσταση δείχνει την κρισιμότητά της και ότι υπάρχουν όλο σύνεχος καινούργια θέματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια με τη συζήτηση. Μια τέτοια συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ. Θέλουμε να είμαστε αποφασιστικοί γύρω από την χρησιμότητα της Agenda 2020 με τόσα εκατομμύρια ανέργους και με 100, εκατομμύρια κόσμο στα όρια της φτώχειας σε μία από τις πιο πλούσιες περιοχές του πλανήτη. Λοιπόν, θα συνεχίσετε τον αγώνα και θα μας δώσετε επιχειρήματα, δεδομένα και θα βοηθήσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σα ευχαριστώ. Okay, friends, uh, now we'll proceed uh, with the uh, number point four on the agenda. Να προχωρήσουμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης ε, που έχει να κάνει με ε, το progress, το χρηματοπιστωτικό μέσω μικροχρηματοδοτήσεων. Και Είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερομένους στις 7 Μαΐου και σήμερα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σούλτσε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα επόμενα λεπτά θα συζητήσουμε το Progress που είναι μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων. Θα θυμάστε ότι το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Ε, αξιολόγησα λοιπόν ε, ενδιαμέσως ε, την αποτελεσματικότητα του μέσου αυτού. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στους άνεργους και τους μειονεκτούντες σε πιστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κλήθηκαν ε, να λύσουν το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότησης των ανθρώπων αυτών. Όσοι ήσασταν παρόντες θα θυμάστε κατά την τελευταία θητεία ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2010 με 250, 205 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας ε, υιοθετήθηκε τον ε, Σεπτέμβριο του 2013 και τέθηκε σε νέα οικονομική βάση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Κομισιόν ε, προβλέπουν ότι το μέσο θα λειτουργήσει έως το 2016. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν, ο μηχανισμός αυτός ε, λειτουργεί πολύ καλά και αντιστοιχεί ε, στους στόχους ε, της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων, το αυτό που δηλαδή μόλις συζητήσαμε. Πολλές θέσεις εργασίας υπάρχουν σε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, και βοηθάει ο μηχανισμός αυτός σε τη δημιουργία και την διατήρηση τέτοιων επιχειρήσεων με την παροχή μικροδανείων. Για τους φορολογούμενους είναι πολύτιμο το μέσο αυτό. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία μικρή επιχείρηση και αυτό είναι καλύτερο από το να του παρέχεται επίδομα ανέργειας για παράδειγμα. Η χρηματοδότηση από το Προγκρέσ επιτρέπει να δίδονται δάνεια σε ανθρώπους ε, που κινδυνεύουν να ε, αποκλειστούν από την αγορά εργασίας. Ο κίνδυνος ε, είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι με συνηθισμένα δάνεια και παρέχεται ο μηχανισμός αυτός σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη. Το γεγονός ότι δεν παρέχεται σε όλα τα κράτη-μέλη οφείλεται σε ε, διαφορετικούς ε, βαθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Καλούνται τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν ακόμα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία. 13.272 ε, δάνεια δόθηκαν και αυτό απέχει λίγο από τον στόχο που είχαμε θέσει. Όσον αφορά την ομάδα στόχο μπορώ να σας πω το εξής, ότι πάνω από το μισό των ε, δικαιούχων δεν θα μπορούσαν να λάβουν δάνειο από ε, τράπεζα. Το 43% βρίσκονται κάτω από το εθνικό όριο της στόχιας, ε, το 17% αυτοχαρακτηρίστηκαν χαρακτηρίστηκαν ως άποροι. Όσον αφορά τις γυναίκες, το ποσοστό γυναικών πιστεύω ότι είναι ευχάριστα υψηλό, το 37% των ε, δικαιούχων ε, είναι γυναίκες. Ε, δεν φτάσαμε το στόχο των 40% που θέλαμε, αλλά τον πλησιάσαμε πολύ. Κάποια αρνητικά συμπεράσματα ότι πολλοί δικαιούχοι λόγω του φόβου να ταυτιστούν με κάποια μειονότητα δεν λένε ότι προέρχονται από μία τέτοια, κάτι που ε, σημαίνει ότι στις στατιστικές δεν φαίνεται ότι ε, έχουν δοθεί πολλές επιστώσεις ε, στις ομάδες αυτές. Καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις βελτίωσης του μηχανισμού. Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας δεν ε, λαμβάνουν εύκολα χρηματοδότηση. Ε, ο ε, ευρωπαϊκός ορισμός των μικροπιστώσεων σημαίνει ότι προβλέπει να βρίσκονται κάτω από 25.000 ευρώ τα δάνεια αυτά. Καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει Ε, μήπως ε, θα μπορέσει να βελτιωθεί η παροχή δανείων ε, προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να στηριχθούν πολύ καλά και ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για αυτές τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό στο μέλλον. Ελλείψεις και προτάσεις βελτίωσης. Σημαντική έλλειψη είναι ότι δεν, δεν προβλέπεται άσκηση των δικαιούχων. Δεν προβλέπεται δηλαδή υποστήριξη όσον αφορά τις λογιστικές εργασίες, για παράδειγμα. Κατά την μικροχρηματοδότηση μας ενδιαφέρει όχι μόνο η οικονομική υποστήριξη, αλλά και η υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων και τις ε, λογιστικές εργασίες. Θα πρέπει ε, και αυτό να επιληθεί στο μέλλον. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ε, που έχουν ωφεληθεί από το Progress θα πρέπει να παρακολουθούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις επιχειρήσεις αυτές και όσον αφορά τον ορισμό της μικροχρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου είναι ξεπερασμένος ο ορισμός αυτός και θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος. Η μικροχρηματοδότηση σύμφωνα με τον ορισμό ε, δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα 25.000 ευρώ και προβλέπεται για ε, επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 πρόσωπα. Ειδικά στην, ε, στη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ χαμηλά τα όρια αυτά. Θα πρέπει να γίνει επίσης σύνδεση με άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι θέσεις μας διαφέρουν από αυτές άλλων επιτροπών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντικό είναι να υπάρχει ευρύτερη χρηματοδότηση για το Progress. Θετικό είναι σήμερα ότι οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πρόγραμμα Progress και το στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ε, υπάρχει διαχειριστής ε, που βοηθάει ε, την διεξοδική του προγράμματος. Και φτάνω στο συμπέρασμα μου. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα μέσο κοινωνικής πολιτικής που βοηθάει ανθρώπους από το περιθώριο της κοινωνίας να ενταχθούν σε αυτήν και να διασφαλίσουν μέτρα διαβίωσης. Θα ήθελα να σας θυμίσω τον Οντάβιο Πίντο, κάποιον δικαιωγό μικροχρηματοδότησης εδώ στο Βέλγιο, που έχει αποπληρώσει τη μικροχρηματοδότηση που έλαβε και έχει αναπτύξει την επιχείρησή του. Σημαντικό όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις είναι να συνδυάσουμε τα δάνεια με κατάρτιση ώστε οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Προσλέπω στην καλή συνεργασία μαζί σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μαζί να βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό. Προσλέπω στην καλή συνεργασία όχι μόνο με τους κοιόδης ε, εισηγητές, αλλά και με τους άλλους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον ε, Χαβιέ Ευχαριστώ. Πράγματι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο εισηγητής είναι τεκμηριωμένη, λεπτομερής και με συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος. Με συγκεκριμένες τροπολογίες νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε κάποια σημεία, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πλήρης ως έχει. Η προσπάθειά μας είναι οι τροπολογίες αυτές να ανοίγουν ακριβώς αυτή την τριπλή προοπτική που πρέπει να έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή απασχόληση, θέσεις απασχόλησης, δεύτερη διάσταση είναι μια διάσταση στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών και τρίτο είναι ένα οικονομικό κίνητρο το οποίο να ανοίγει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο μέσα από παραδοσιακά, από παραδοσιακούς τρόπους δεν μπορεί να επιτευχθεί. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μικροχρηματοδότησης στα πλαίσια και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για επενδύσεις θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ακριβώς τις κοινωνικές ε, ε, επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρξουν από την εφαρμογή του προγράμματος αυτούς και να μην ξεχάσουμε την διάσταση του φύλου εδώ έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να συνεχίσουμε να, για να πετύχουμε ένα θετικό βήμα. Να εξετάσουμε επίσης την δυνατότητα να συμπεριλάβουμε και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ή κάποιες άτυπες οικονομικές μορφές. Και τέλος εμείς συμμεριζόμαστε για τον τρόπο ενίσχυσης ακριβώς της μαθητείας και της κατάρτισης για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη από μικροπιστώσεις Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο παραδοσιακό πιστοτικό σύστημα και στο συγκεκριμένο. Το θέμα είναι όπως είπαμε να προσπαθήσουμε να το καταστήσουμε πιο διαθέσιο, να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με, με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Τεμπέσιους, εκπρόσωπος της ομάδας των συντηρητικών. Χωρίς μικρόφωνο. Με ακούτε τώρα. Κύριε εισηγητά θα επαναλάβω σύντομα αυτά που είπα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την έκθεσή σας είναι πολύ πλήρης και ήδη αναφερθήκατε σε πολλές στοιχείες του θέματος. Ευχαριστώ. Επίσης περιγράψατε πολύ καλά τα διάφορα προβλήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα που θα θέλαμε να συμπληρώσουμε. Καταρχάς έχουμε το ρόλο των τραπεζών. Εάν θέλουμε να δίνουμε κρατικά δάνεια, το πρώτο ερώτημα είναι γιατί να το κάνουμε αυτό. Συχνά η απάντηση είναι ότι υπάρχουν εδώ ελλείψεις στην αγορά. Είναι αλήθεια αυτό. Κάποιες τράπεζες στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν πολύ χαμηλά ίδια κεφάλαια για να παρέχουν ε, δάνεια. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει εδώ αποτελεσματικός ε, τραπεζικός τομέας ε, και γι' αυτό θα πρέπει η πολιτική να ασχοληθεί με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και να καλύψει το κενό. Αντί γι' αυτό όμως υπάρχουν διάφοροι ε, μηχανισμοί ε, μεταφοράς ε, κεφαλαίων που απλά καταπολεμούν τα συμπτώματα. Το 17% των δανειοληπτών είχαν απορριφθεί από εμπορικές τράπεζες, είπατε και πολλοί υπέβαλαν αίτηση επειδή θεώρησαν ότι θα τους απέριπτε μια, μια τράπεζα. Ε, δεν μπορούμε όμως να δημιουργούμε ένα μέσο για τους ανθρώπους ε, που απλά δεν κάναν τον κόπο να κάνουν ε, αίτηση σε κανονική τράπεζα. Επίσης δεν θα πρέπει να περιοθωριοποιήσουμε την ιδιωτική οικονομία. Στις κάτω χώρες υπάρχει ένα σύστημα όπου πρόσβαση στις κρατικές μικροχρηματοδοτήσεις έχουν μόνο όσοι ήδη έχουν απορριφθεί από εμπορικές τράπεζες. Επίσης, όσον αφορά την ε, κατάρτιση και την παρακολούθηση, κατά τη γνώμη μου είναι επίσης ε, σημαντικό να στηρίξουμε τους συμμετέχοντες ε, με προγράμματα κατάρτισης. Συμφωνώ δηλαδή με τη θέση του εισηγητή, θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί το κόστος αυτό να το φέρει το ίδιο το πρόγραμμα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για άλλες ε, δαπάνες του προγράμματος αυτού. Τρίτον, ε, θέλουμε εμπειρική παρακολούθηση του προγράμματος. Ε, σημαντικό είναι αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν εδώ διάφορες πτυχές. Για παράδειγμα, τα ποσοστά επιτυχίας ε, θα πρέπει ε, να αναλυθούν ε, ανάλογα με τις μειονότητες, την ηλικία, το φύλλο κλπ. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό οι γυναίκες να έχουν πολύ καλό ε, ποσοστό αποπληρωμής ε, με βάση την εμπειρία που έχουμε από άλλα προγράμματα. Αυτές λοιπόν ε, θα είναι και πιο ελκυστικές για τις εμπορικές τράπεζες. Επίσης, όσοι έχουν εγκαταλείψει το πρόγραμμα, πώς τα πήγαν και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτό. Προσβλέπω στην καλή μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιωβα, που εκπροσωπεί τους φιλελεύθερους. Πολύ λίγα σχόλια. Ε, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία. Η κυρία Ρενάτα Βέμπερ βλέπει μία κοινή προσέγγιση ε, ως προς το πρόγκρες στην μικροχρηματοδότηση. Η Ρενάτε θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία για να ε, βοηθήσουμε την, ε, στην κεφαλαιοποίηση των ευρημάτων αυτής της έκθεσης και επειδή συμμετέχω και στην Επιτροπή Κοντ θα ήθελα να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα εκπονήσει μία έκθεση για την μικροχρηματοδότηση μέχρι τα τέλη του Ιουνίου και νομίζω ότι θα έχουμε μία συνολική εικόνα για το πώς λειτουργεί η μικροχρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ από τους φιλελεύθερους. Ε, από την εκπρόσωπος δεν είναι εδώ. Ε, ε, από τους πράσινους σκιώδης. Ε, δεν είναι παρούσα. Ούτε η κυρία Λάμπερτ. Ε, ζητάτε το λόγο μετά τους σκιώδης. Η κυρία Πέκκινη που εκπροσωπεί το FTD. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την έκθεση που είναι άκρος ενδιαφέρουσα και μας δίνει δεδομένα που δεν γνωρίζουμε όλοι. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία διάρθρωση μικροχρηματοδότησης, δεν το γνωρίζουν όλοι. Θέλουμε να φτάσουμε σε 46.000 μικροχρηματοδοτήσεις μέσα στα πλαίσια των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, έχουν ήδη ε, εκδοθεί μικροχρηματοδοτήσεις σε 152, άρα εκλείπει ένα 95%. Υπάρχει όμως η θέληση και η ζήτηση. Βέβαια, η ζήτηση είναι πολύ υψηλότερη από την προσφορά. Αυτά τα μέσα χρειαζόμαστε και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν ε, ε, πολλοί απραγματοποιητοί, θα μπορούσαν να πω, ε, πολλαπλασιαστές σαν αυτούς που προτείνει το σχέδιο Juncker. Θα πρέπει να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη και από τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί το 85% αφορούν μικροεπιχειρήσεις. Οι μικροεπιχειρηματίες όμως ε, δεν ε, έχουν πάντα πρόσβαση στις δανειοδοτήσεις, διότι αποτελούν ε, μία μειοψηφία για τα τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με, την ευρωπαϊκή, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις που αποσχολούν κάτω από 10 εργαζόμενους, ίσως και αυτός ο ορισμός θα έπρεπε να επανεξεταστεί. Μιλάμε λοιπόν για κοινωνική πολιτική, πολιτική. Η έκδοση αυτών των πιστώσεων, των δανείων δεν είναι παρά δαπανηρή για τις τράπεζες και θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ καλύτερο να χορηγούνται αυτά τα δάνεια σε σχέση με επιδόματα ανεργίας που θα πρέπει να καταβληθούν. Άρα θα ήταν κάτι το πολύ προσοδοφόρο για τις ΜΜΕ. Ριμπέιρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ε, να συγχαρώ τον κύριο Σούτσε για την έκθεση. Είναι πολύ καλά διαρθρωμένη η έκθεση και επίσης ε, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα λύσεων. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σε κάτι και είναι το εξής. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να επιληθεί το ζήτημα. Είναι ένα μέσο κοινωνικής πολιτικής και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι μικροπιστώσεις αφορούν κυρίως ανέργους. Δηλαδή, αν δεν είχαν πρόσβαση στα μικροδάνεια αυτά, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Από ό,τι είδα ε, υπάρχει παραπλάνηση και παραπληροφόρηση στα κράτη-μέλη. Δηλαδή πέρα από το πρόγραμμα που πρότεινε ο κύριος Σούτς και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να προωθήσουμε την πληροφόρηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων και των ανέργων. Θα πρότεινα λοιπόν και θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση να αποτανθούμε στους οργανισμούς ανέβρες εργασίας, στα πανεπιστήμια και στα εθνικά ιδρύματα τα οποία προβάλλουν πρωτοβουλίες για τις μικροεπιχειρήσεις καθώς και στα εμπορικά επιμελητήρια έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλο ένα και περισσότεροι πολίτες σε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, deadline. Σας ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 15η Σεπτεμβρίου η εξέταση των τροπολογιών 12 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου η υιοθέτηση των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο 5. Ανταγωνιστική αγορά εργασίας για τον 21ο αιώνα. Αντιστήχηση ικανοτήτων και αναγκών. Έχει το λόγο η συγγήτρια. Θα είμαι συντομότερη από ότι ο τίτλος της έκθεσής μου. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες, 360 περίπου. Είχαμε μία πρώτη συνάντηση των σκιωδών που κράτησε τρεις ώρες την προηγούμενη εβδομάδα και συζητήσαμε τις τροπολογίες αυτές, τις ομοιότητές τους και τις διαφορές τους. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν γενικά θετικό. Στόχος είναι να έχουμε το κείμενο απλό, ξεκάθαρο και να μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές μήνυμα μέσω της έκθεσης αυτής γύρω από το τι θέλουμε να μεταφέρουμε. Θα πρέπει στα πλαίσια των συμβιβαστικών προτάσεων να κρατήσουμε τους αρχικούς στόχους και να διασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει για μένα τρεις βασικούς στόχους. Πρώτος, πρέπει να αντιστοιχίσουμε καλύτερα τις επαγγελματικές ικανότητες και τις ανάγκες της αγοράς να προβλέψουμε τις ανάγκες για το μέλλον, να συνεργαστούμε στενότερα σε επίπεδο οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Δεύτερη προτεραιότητα και δεύτερη στόχος είναι να προτείνουμε κάποιες, κάποια βήματα για μεγαλύτερες μορφές συνέργειας, να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ηλικίες, και εδώ φυσικά και τους μεγάλης ηλικίας εργαζομένους. Και τρίτος στόχος είναι να μάθουμε και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαιτείται μία συνταγή για όλους, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους. Είμαι υπέρ των τροπολογιών λοιπόν που δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα από την αρχική πρόταση. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια απλή και συνοπτική πρόταση. Θα προτείνω συμβιβαστικές τροπολογίες όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τροπολογίες οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της έκθεσης. Ελπίζω ότι θα υπάρξει απαιτούμενη συνένεση και θα συμφωνήσουμε στο περιεχόμενο. Αύριο το απόγευμα έχουμε άλλη μία συνάντηση Νομίζω ότι ακολουθούμε την σωστή κατεύθυνση. Να ακούσω λοιπόν τώρα τις απόψεις και των άλλων πολιτικών ομάδων και τις ε, εντυπώσεις που έχουν από την προηγούμενη, αν και δεν είναι εδώ παρόντες ε, όλοι οι σκιώδεις, είναι Δευτέρα απόγευμα και πολλές είναι οι πτήσεις που έχουν καθυστερήσει σήμερα. Εν πάση περιπτώσει περιμένω τα σχόλια των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστούμε. Ακούμε ότι η κυρία Γιασλοβιάκα θα φτάσει πριν τελειώσει η συνεδρίαση. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο του σκιώδους εισηγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Γιονκύριος δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Ευχαριστεί για την έκθεση αυτή η οποία περιέχει κάποια σημαντικά στοιχεία. Δεν δίνει όμως συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας διότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στις δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα και την ανεξαρτησία. οι συντάξει, τα συστάματα κοινωνικής ε, ασφάλισης ε, ε, δεν αναφέρονται επαρκώς. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα κριτήρια, θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και πιο βιώσιμες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας όλα αυτά να προκύπτουν σαφώς από την έκθεση αυτή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση και με τις θέσεις ασκούμενων που να παρέχουν ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Πολλοί νέοι ε, έχουν άμυστες θέσεις ασκουμένων, οι οποίες όμως ε, εξωθούν ε, τους μισθωτούς εργαζομένους. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι χρειαζόμαστε ένα ποιοτικό πλαίσιο για αυτές τις θέσεις. Στην έκθεση αναφέρεται η κινητικότητα των νέων εργαζομένων, απαιτείται μάλλον θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η κινητικότητα θα πρέπει να είναι ποιοτική και όχι να εξυπηρετεί την μείωση των αμοιβών. Θα πρέπει να είναι εθελοντική κινητικότητα και θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση ότι αντιμετωπίζουμε δημογραφικές εξελίξεις Πιστεύω όμως γενικά ότι η έκθεση αυτή επικεντρώνεται υπερβολικά στο ότι οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά ε, επειδή δεν ε, έχουν αρκετά κίνητρα. Αυτό είναι λάθος. Το θέμα δεν είναι τα κίνητρα και οι κυρώσεις. Ε, θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αποδιδεγμένα καλές πρακτικές. Σωστή διαδικασία δεν είναι η πολιτική λιτότητα σε, σε κάποιες χώρες. Ακριβώς έχουν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης με κρατικές επενδύσεις και αυτό είναι μια πρακτική που έχει αποδείξει την αξία της. Αυτά από μένα. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε αρκετή δουλειά για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες πάντως έχουμε πολύ σαφή εικόνα του τι θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς από το ECR? Όχι. Από την ΚΟΕ? E? Όχι. Θα δώσω το λόγο στον Τέρι και από τους Πράσινους. Ε, thank also. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και πόσο πιστεύουν, πόσοι πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το θέμα είναι ζωτική σημασίας για τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπε η Γιούτα Στάινρουκ. Δεν θα πρέπει να δώσουμε την εικόνα των ε, άνω των 5 εκατομμυρίων ε, ανέργων στην Ευρώπη, ότι είναι άνεργοι δηλαδή, γιατί δεν προσπαθούν αρκετά. Αυτό αποστέλει το λανθασμένο μήνυμα προς τους ε, νέους, που προσπαθούν, έχουν πολλές δεξιότητες, πολλά προσόντα, αλλά δεν βρίσκουν εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σταλεί το μήνυμα ότι, το μήνυμα ότι τα προσόντα ε, ενισχύουν τις δυνατότητες αυτών που θέλουν, θέλουν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Η χρήση των βέλτιστων πρακτικών είναι ύψης της σημασίας για να επιλύσουμε ε, αυτά τα επιμέρους ζητήματα τα οποία δημιουργούν διχογνωμίες. Καταρχήν, ως προς τα κίνητρα για εργασία, εμείς ως πράσινοι πιστεύουμε ότι τα κίνητρα δίνονται όχι πιέζοντας τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, και μη ε, αναφέροντας την ασυμετρία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ή εργαζομένων και ανέργων, αλλά ενισχύοντας τους ανέργους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και για να μπορέσουν να έχουν καλή ποιότητα ζωής και να έχουν και κοινωνική προστασία. Το δεύτερο ζήτημα είναι η συμμετοχή οργανώσεων ε, που ασχολούνται με θέματα ανεργίας και έχουν πληγεί από την ανεργία και που ακριβώς θέλουν να έχουν ε, κοινωνική προστασία, δηλαδή μετανάστες, γυναίκες και φοιτητές που θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Και ένα άλλο θέμα, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες είναι κάτι που σχετίζεται άμεσα με την αγορά εργασίας, αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε αυτό το διεξοδικό ε, χαρακτήρα, γιατί οι δεξιότητες βοηθούν και η εκπαίδευση αφεαυτής. Γι' αυτό μιλάμε και για την προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων όλων των ηλικιών θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι έναν ευρύτερο ορίζοντα της ε, κοινωνίας στην οποία ζουν. Αυτή είναι μία από τις διαστάσεις της δημοκρατίας και θα θέλαμε και η εκπαίδευση να ενταχθεί σε αυτή την έκθεση. Προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση, γνωρίζω τα θέματα που μπορούν να οδηγήσουν σε διαφωνία, αλλά πιστεύω ότι επικοδομητικά μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα επιμέρους ζητήματα. Ευχαριστώ. Λάουρα, Άγγια, θέλετε το λόγο και κυρία ε, Μπέγκιν. Εγώ θα προσπαθήσουμε να συνοηθούμε. Έχει υπάρξει μια παρανόηση, λέει η κυρία Μπεγκίν. Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας. Είχαμε μια καλή συζήτηση στα πλαίσια της συνάντησης των σκιωδών έχει μεγάλη σημασία να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας και να αντιστοιχεί η ζήτηση με την προσφορά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Το θέμα δεν είναι μόνο κατανομή πόρων, αλλά δυστυχώς έλλειψη θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ με τις συμβιβαστικές προτάσεις που εν πολλής είναι δεκτές, κάποιες μόνο μορφές σχολείων, σχολείων για το ότι οι πολιτικές λιτότητας έχουν χειροτερεύσει την οικονομική κρίση και στην Ευρώπη και συνεχίζονται και επαναλαμβάνονται οι πολιτικές αυτές, εμείς θα καταθέσουμε μια τροπολογία. Και σχετικά με τη συμβιβαστική F αγγλικό, εμείς δεν συμφωνούμε με το ότι θα πρέπει ε, ο πολίτης να εργάζεται περισσότερα χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με ένα πληθυσμό μεν που γυράσκει, αλλά η παραμονή στην αγορά εργασίας μακροπρόθεσμα στην παρούσα φάση δεν έχει λογική. Θα πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά η πρόταση αυτή λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλύτερη θέση για αυτούς που χάνουν την εργασία τους σε ένα σημερινό οικονομικό πλαίσιο για το H αγγλικό. Όπως είπε ήδη η σκιώδης της Γκουε και εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω πλήρως την ιδέα ότι δεν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Νομίζω ότι ε, δεν ε, εργάζονται ορισμένοι ότι δεν θέλουν, αυτό δεν ισχύει. Σε μια χώρα σαν τη δική μου όπου η ανεργία είναι 12% και των νέων είναι πάνω από απίστευτα ποσοστά, το θέμα είναι να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χώρες. Θέλουμε λοιπόν μια διατύπωση λίγο διαφορετική αν και κατανοώ την ιδέα η οποία λέει ότι θα πρέπει ε, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε με πιο εύκολο τρόπο την πρόταση. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην κινητικότητα αλλά δεν θα πρέπει να είναι κάτι το υποχρεωτικό και δεν είναι αποκλειστικά μέσο θα έλεγα για την καταπολέμηση της ανεργίας και νομίζω ότι στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών ε, θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καταφέραμε λοιπόν να περιμένουμε για την κυρία Γιασλοβιέσκα η οποία είχε προβλήματα όπως και πολλοί από εμά σήμερα με τις πτήσεις της. Θα σας ακούσουμε σαν σκιώδη εισηγήτρια του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Λαμπάγιοβα. Αυτά τα οποία μας είπε έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης οι οποίες δεν καλύπτονται σε ορισμένες χώρες γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Ή πολλές φορές οι θέσεις αυτές δεν είναι γνωστές. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα που δεν ακολουθούν α, κάποιες διαδικασίες κατάρτισης, δεν κάνουν στάζ και η έκθεση αυτή σε αυτούς απευθύνεται έτσι ώστε να ενδιαφερθούν και με διαφορετικό τρόπο για το μέλλον τους. Πόσο μάλλον που σήμερα η αγορά εργασίας είναι πολύ δύσκολη για τους νέους και για αυτούς που είναι άνω των 50 επίσης. Πολύ συχνά ακούμε ότι αυτοί που είναι άνω των 50 δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εργαστούν. Η έκθεση αυτή έχει προκαλέσει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον, όπως δείχνουν οι 360 τροπολογίες, πρόκειται για προτάσεις πολύ ενδιαφέρουσες και επ' αυτής της βάσεως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια <clears throat> θετική έκθεση για όλους. Όλα θα εξαρτηθούν φυσικά από την ε, εισηγήτρια, αυτή θα μας προτείνει την τελική διατύπωση. Υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά ε, στοιχεία κατανοητά θα έλεγα και για τα κρατημέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως για τους στόχους αυτής της πρότασης. Νομίζω ότι μια ανταγωνιστική αγορά στην Ευρώπη είναι βασικός στόχος για την επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση ε, του επίπεδου της αγοράς εργασίας με συγκεκριμένες μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ε, ικανότητες και γνώσεις. Πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές όπου αυτές είναι υπεύθυνε για θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης την επιχειρηματικότητα, να επενδύσουμε στην κατάρτιση και των εργοδοτών γιατί όλο και περισσότερο βλέπουμε να υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι σε αυτήν την περίοδο κρίσης χρειάστηκε να απολύσουν. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω εδώ άλλες και δεν χρησιμοποιούν εδώ άλλες δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους όπως να επενδύσουν στους ίδιους τους εργαζομένους τους. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει η δυνατότητα εδώ να αναγνωρίσουμε και τους εργαζομένους που έχουν την ικανότητα για μια συγκεκριμένη θέση απασχόλησης, αλλά η θέση αυτή ε, δεν έχει διάρκεια. Θα πρέπει να εμείνουμε στην κατάρτιση των νέων για να καταστούν υπεύθυνοι για το μέλλον τους, για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με μεταρρυθμίσεις της εργασίας, έτσι ώστε ε, να γίνουν όλοι δραστήριοι και να αντιδράσουν γρήγορα στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την Λαμπάχοβα για την εξαιρετική της έκθεση. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που κατέθεσαν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μάκιντάιρ. Λυπάμαι που δεν ήμουν στην αρχή αυτή της συζήτηση, αλλά είχαμε πρόβλημα να φτάσουμε σήμερα. Ελπίζω, χαίρομαι μάλλον, που έφτασα για να μπορέσω να κάνω ορισμένα σχόλια. Η Μαρτίνα έχει επιτελέσει εξαιρετική εργασία, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και μπόρεσε να συμπεριλάβει όλα όσα μας απασχολούν. Μιλάμε για ευέλικτη αγορά εργασίας, για την ανάγκη αυτής και αυτά τα συζητήσαμε μεταξύ όλων των σκιωδών πώς μπορούμε να έχουμε την υποστήριξη ολόκληρου του πολιτικού φάσματος. Αυτό που έχει σημασία είναι να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες και Μιλάμε για ε, επιχειρηματικές δεξιότητες των νέων ανθρώπων για να μπορέσουν να γίνουν επιχειρηματίες και όχι μόνο ε, εργαζόμενοι αλλά και εργοδότες. Ως προς τις δεξιότητες θα ήθελα να συγκεντρωθούμε στην ανάγκη της μαθητείας ε, δεν χρειάζεται όλοι να αποκτήσουν δεξιότητες από τα πανεπιστήμια. Μπορούμε και από την επαγγελματική κατάρτιση να τις αποκτήσουμε ή από τα συστήματα μαθητείας που βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να ενώσουν περισσότερο την εκπαίδευση με την εργασία. Μιλήσαμε για 361 τροπολογίες και είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση σκιωδών την προηγούμενη εβδομάδα όπου είδαμε όλες τις προτάσεις συμβιβασμού που καταρτίστηκαν. Πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν δύο προτάσεις συμβιβασμού που δεν με βρήκαν σύμφωνοι, απόλυτα σύμφωνοι, αλλιώς μπορώ να ε, δεχτώ τις περισσότερες. Όλοι συμφωνήσαμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις. Δεν είναι εύκολο για την εισηγήτρια, αλλά αυτό γνωρίζω ότι θέλει να το κάνει η Μαρτίνα. Γι' αυτό θα ήθελα να μην υπάρχουν επαναλήψεις να μην έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά μια σαφή έκθεση που να εστιάζει την προσοχή της στα βασικά ζητήματα. Νομίζω ότι όλες οι ιδέες είναι σημαντικές, και θα πρέπει να μας καθοδηγήσει για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε τις ευκαιρίες για να αποκτήσουν ε, οι άνθρωποι εργασία. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική έκθεση, η έκθεση και ελπίζω η Επιτροπή να τη λάβει υπόψη και να καταρτήσει πολιτικές υποστηρίζοντας αυτές τις ιδέες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τη Μαρτίνα και προσμένουμε την επόμενη συνάντηση των σκιωδών για να φτάσουμε σε, περαιτέρω συμβιβασμούς. Η κυρία από το EFTD. Ευχαριστώ. Η έκθεση αναφέρεται στην κινητικότητα των εργαζομένων και θα ήθελα να πω ε, ε, καλύτερα να μιλάτε για την ανοιχτή μετανάστευση. Θέλουμε ένα αυστραλιανό σύστημα, δηλαδή ε, άδειες παραμονής με βάση τις δεξιότητες. Στην παράγραφο 23 μιλάμε για εργαζόμενους με προσόντα από τρίτες χώρες. Ο κύριος Κάμερον είπε ότι ίσως φτάσουμε και σε ε, και σε απόκτηση εργασίας από Ινδούς και αυτό αφορά, μπορεί να αφορά μέχρι ε, ένα πολύ υψηλό αριθμό εργαζομένων που θα θέλουν βέβαια και ένα σύστημα πρόνοιας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει αυτό το άνοιγμα το οποίο προσελκύει εργαζόμενους από τρίτες χώρες ε, πλημμυρίζοντας, δημιουργώντας μια πλημμυρίδα εργαζομένων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να τονίσω τις ε, τροπολογίες 2, 2, και 4 3-4, ε, μιλώντας για ελάχιστο μισθό. Πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ε, μισθών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς ε, μπορείτε να φτάσετε σε αυτό το υπερκράτος που θέλετε. Μα δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να προωθείτε νομοθεσία, τέτοια νομοθεσία. Θα ήταν ε, η οικονομική καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει έναν κατώτερο μισθό. Η κυρία Λαμαγιώβα. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική συζήτηση. Λέει η κυρία Νταβαγιώβα, αλλά θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε και σε μία ε, φιλοσοφική συλλογιστική για την αντιμετώπιση του θέματος. Ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και φιλοσοφικά ακόμα το ζήτημα για τα κίνητρα των νέων, την ευθύνη για την τύχη τους. Μιλήσαμε και για τη σύνταξη του κειμένου, πώς λέξεις σε συγκεκριμένη γλώσσα έχουν διαφορετική εντελώς σημασία. Η, τι σημαίνει ευθύνη όταν μιλάμε για ευθύνη στην έκθεση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα και ευχαριστώ του Σκιώδης. Τώρα ε, θα ασχοληθούμε με τους νέους συμβιβασμούς, θα τους αποστείλουμε αμέσως μετά την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής και θα ήθελα να πω ότι πολλά ζητήματα έχουν αλλάξει γιατί ε, τα είδαμε ήδη στη, στους και γι' αυτό ακριβώς θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Διαβάστε τους νέους συμβασμούς πριν, πριν από αύριο. Αύριο έχουμε τη συνάντηση των σκιωδών και ίσως θα ήταν σκόπιμο να δείτε αυτούς τους συμβασμούς πριν προτείνετε νέες τροπολογίες γιατί έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Ε, κάτι το πολύ σημαντικό που τονίστηκε και το είπα στην αρχή Νομίζω ότι ο στόχος είναι να κρατήσουμε το κείμενο όσο πιο απλό και σαφές γίνεται. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις επαναλήψεις, να αποστείλουμε σαφή μηνύματα και να μιλήσουμε πραγματικά για δεξιότητες και προσόντα. Να μην κάνουμε έναν συνονθήλευμα δηλαδή γιατί βεβαίως υπάρχει το δέλεαρ να τα συμπεριλάβουμε όλα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα απλό μήνυμα προς όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη εργασία για μας αύριο, αλλά με τη βοήθεια των σκιωδών θα τα καταφέρουμε. Και αν σας ενδιαφέρουν οι φιλοσοφικές ε, μας συζητήσεις, μπορούμε να σας δώσουμε ορισμένα στοιχεία την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα. Μιλώ για τους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ. Στις 23 Ιουνίου θα εγκρίνουμε την έκθεση στην Επίτροπη. Αυτά έχουμε να πούμε. Αυτό ήταν και το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε κιόλας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ευχαριστώ. Γεια σας.